Αγαπητοί συνάδελφοι, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Και προχωρώ στο επόμενο σημείο στη μέση διάταξη που είναι η έκθεση σε σχέση με τις συνεδρίες των συντονιστών. για τους εισηγητές. Η πρόταση κανονισμού που θεσπίζει ε, ένα πλαίσιο για, τα, για την πρόσβαση σε λιμενικές υπηρεσίες είναι η ομάδα των σοσιαλιστών που θα αναλάβει το θέμα αυτό, δεύτερη έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας 32 του 2000 για τις τεχνικές τεχνικούς ελέγχους ε, στην ε, άκρη των δρόμων δεν θα υπάρξει καμία δράση από τη δική μας πλευρά. Υπήρξε μία αγρομοδότηση τώρα σε σχέση με την ε, διαχείριση, οικονομική διαχείριση στην περίπτωση χωρών, στην δημοσιονομική διαχείριση για χώρες που έχουν σοβαρές δυσκολίες, καμία δράση, για τα έγγραφα για πληροφόρηση η ανακοίνωση για τους λιμένες θα συνδεθεί με την προηγούμενη εκθέση που αναφέραμε. Το ίδιο με την στρατηγική για την κλιματική αλλαγή. Γιατί ούτε εκεί απλά κάνουμε τίποτα. Συμφώνησαν οι συντονιστές για το σχέδιο επιστολής που θα στείλουμε σε σχέση με τους κανόνες βάσει του άρθρου 49 για τους επιβάτες αεροπορικών εταιριών και έτσι η ΙΜΚΟ μπορεί να συμμετάσχει στις συζητήσεις μας, αλλά δεν έχουν δικαιώματα να συμμετέχουν στον τελικό τριμερή διάλογο. Για την επιστολή της Επιτροπής ΕΚΟΝ που ζήτησε να μπει κάποιος στην ομάδα εργασία για τα θέματα ανταγωνισμού, η πρόταση του ε, η πρόταση είναι να είναι ο κύριος Ρίκε <clears throat> για τις ε, κατεχώρηση πράξης εδώ υπήρξε μια αίτηση από το ΕΛΚ, από το συντονιστή του ΕΛΚ. Η απόφαση είναι ότι η Γραμματεία θα στείλει ένα υπόμνημα για το θέμα αυτό και θα έχουμε μια συζήτηση μεταξύ συντονιστών για τη σημασία των ε, κατεξουσιοδότηση πράξεων στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών. Οι συντονιστές επίσης κατέγραψαν τα ενημερωτικά δελτία 12 και 13 και επίσης για τον περιορισμό των ορών πτήσης είχαμε μια παρουσίαση από τον κύριο Μπόλτουιν από την ε, Γενική Διεύθυνση Μεταφορών της Κομισιόν και έλαβαν γνώση οι συντονιστές αυτής της παρουσίας. Αυτά από τους συντονιστές. Είστε ευτυχισμένοι? Πολύ καλά. Εγκρίνονται λοιπόν όλα αυτά. Ερχόμαστε στο επόμενο σημείο που είναι... Για να μαζέψω τα χαρτιά μου. go to Tintin. Okay, it's now the votes. Ψηφοφορίες τώρα. Η έκθεση για τους ψηφιακούς ταχογράφους. Κυρία Τσίκαου. Εντάξει. Μία δοκιμαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Has everybody voted? Όλοι ψηφίσατε. Πέρας. Is okay, Adi. Εντάξει. Ναι, ναι, ήδη σε έχω υπολογίσει. They don't go over quota on that then. Εντάξει, έχουμε το σωστό αριθμό λοιπόν από τους σοσιαλιστές. Εντάξει. Oh, first one is the... Έχουμε λοιπόν στην αρχή τον κανονισμό που τροποποιεί τον κανονισμό του Συμβουλίου 3281 για τους καταγραφείς της οδηγίας μεταφορές και τον κανονισμό 561 του 2001 για τους ψηφιακούς ε, ταχογράφους. Η κυρία Τικάου είναι ε, αρμόδια. Άρχεται η ψηφοφορία, είναι μονάχα μία ψηφοφορία χωρί τροπολογίε. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. «33 υπέρ, 3 κατά με μία αποχή. Συγχαρητήρια Σίλβια. Ακολουθεί κυρία, η γνωμοδότηση της κυρίας Βίλς. Πρόταση οδηγίας. για καύσιμο ποιότητος, τροποποίηση της οδηγίας παριθμών 28. Πάμε. Τροπολογία 77 Taylor, υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος ηλεκτρονικός για να ξεκινήσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 22 υπέρ, 14 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 78 Τέιλορ υπέρ. Κατά. Αποχές, η ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται στις 79, 80 και 81 που είναι ταυτόσιμες ψήφι υπέρ κατά απόχες απορρίπτονται 82 υπέρ κατά απόχες απορρίπτονται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 88. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 90. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 91. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 93, 94 αλλά και 95 και 96 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 97 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε για την 97 παρακαλώ, άρχεται. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. 22 με 15. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ κατά αποχές, όχι θα ελέγξουμε την 100, ηλεκτρονικός έλεγχος, αρχική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας, απορρίψατε. 17 με 21. Πάμε στην 110. Τεγράντες Πασκουάλ. Εντάξει, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 111, 112, 113 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 4 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 1-1-4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 116 άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος για την 117. Άρχεται. Εγώ λέω ότι εγκρίνεται, αλλά θα το δούμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Πράγματι εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά. 119 πάλι υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 119 Γίτσες κύριε Κουσέρη ψηφίσατε όλοι πέρας Απολύψατε πράγματι όπως σας το είπα Συμβιβαστική 2 Κύριε Έρτογκ, και εσείς με τις υγείας σας. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 7. Νόμιζω ότι εγκρίνεται εξαρτάται από τους πράσινους. Ψηφίσατε όλοι, πέρας, εγκρίθηκε. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε 121. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 147, όχι, όχι, συμβαστική 4 πρώτα. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα είναι 147 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 146 υπέρ, κατά αποχές Έλεγχος για την 146, εγώ νομίζω ότι εγκρίνεται. 146 έλεγχος άρχεται. Ψηφίσατε όλοι, πέρας, εγκρίνεται. 148 <clears throat> υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 149 και 150 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 151 υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος είναι 151 παρακαλώ. Νόμιζα απορρίπτεται. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται όμως. 152 υπέρ. Κατά. Απόχες απορρίπτεται. 153 υπέρ. Κατά. Απόχες απορρίπτεται. 154, 155, 156 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 159 υπέρ κατά άποχες δεκτή. 160 ε, και 161 υπέρ κατά άποχες απορρίπτονται. 10 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. 162-163 εκπίπτουν. Προχωρούμε στην 165. υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 166 υπέρ, κατά, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 173 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 174 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 177, 178, 179, 80, 81 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 182 υπέρ κατά αποχές νομίζω και αυτή απορρίπτεται θα ελέγξουμε την 182 ηλεκτρονικά άρχιτη ψηφοφορία το S&D έχει οι σοσιαλιστές έχουν ένα παραπάνω που ψηφίζει εντάξει ναι. πέρας απορρίπτεται 183-184 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 1, 91. υπέρ. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 12 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε τη 12 παρακαλώ άρχεται ψηφίσατε όλοι πέρας 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 22 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 22 παρακαλώ άρχεται Ψήφισατε όλοι, πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8, υπέρ. Κατά. Αποχές, δεκτή. 31 ένα, υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος πάλι, άρχιδη ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι, πέρας. Εγκρίντ, 32, υπέρ. Κατά. Αποχές, να ελέγξουμε και την 32 παρακαλώ, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 και 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 30 Έλεγχος εντάξει για τη 41, άρχεται η ψηφοφορία. Οι φιλελεύθεροι άλλαξαν άποψη μάλλον. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Α, συγγνώμη, εκπίπτει, εκπίπτει. Πάμε στη 42 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για τη 42, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 43, 44, 45 και 46. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. 48. Υπέρ. Ναι, ναι, απορρίφθηκε είναι. Σωστό. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές έλεγχος Γιατί 52 άρχεται η ψηφοφορία Ψήσατε όλοι πέρας 50, η 50 εκπίπτει. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 57 και 59 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 56. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. απολύτω. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πάλι. Υπέρ. Υπέρ. 55 κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται. σφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στη 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65, 66 και 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72, 73, 74, 75 και 76 ψήφι περ κατά, αποχές, έλεγχος. Νομίζω ότι εγκρίνονται, αλλά άρχεται η ψηφοφορία για αυτή την πεντάδα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Και πράγματι εγκρίνονται. 20-19. Τελευταία λουκούμια ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 32 υπέρ 6 κατά μία αποχή εγκρίνεται συγχαρητήρια στην κυρία Βίλς. Επόμενη γνωμοδότηση του κυρίου Κράμερ. Δίνω μια έκθεση. Είστε έτοιμοι. Let me just get all my papers in place here τακτοποιήσω λίγο τα χαρτιά μου. Ξεκινούμε με την ε, τροπολογία 8 της κυρίας Μπιλμπάου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά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 αποχές εγκρίνεται, 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 21 υπέρ, κατά, αποχές. Ε, παλήθευση για την 21 παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, Πέρα της ψηφοφορίας, απορρίπτεται ε, λόγω ισοψηφίας. 23 υπέρ, κατά, αποχές, Επαλήθευση για την 23, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. 23, πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση για την 24 παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται, λόγω ισοψηφίας και πάλι, 25 υπέρ, κατά, άποχες επαλήθευση και για αυτή. Αν δεν κάνω λάθος το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουμε, αλλά άρχεται η ψηφοφορία παρόλα αυτά. Ψήφισαν όλοι, πέρασε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία α, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν στη Ρέτζη 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκριμήματα στη Ρέτζη 5. Υπέρ. Σε δύο τμήματα, υπέρ για το πρώτο τμήμα, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τριάντα. Συγγνώμη, αλλά χάλασε το μηχάνισμα ψηφοφορία των σοσιαλιστών. 30. Το του κυρίου Λιμπεράτσκι, υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. 33 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. απόχέ, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα έχει νόημα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Του κυρίου Ντεμπάκερ επειδή ε, κατέπεσε υπέρ, κατά, αποχές, να κάνουμε μια επαλήθευση για την 32 παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 στη συνέχεια ως προστίκη. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική γάμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 44 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση για τη 49, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται λόγω ισοψηφία. 50. Της κυρία Τσικάου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51. Υπάρχει προφορική τροπολογία του κυρίου Κράμερ, ο οποίος προσθέτει end intermodality. Υπάρχει ένσταση. Αν όχι, ψηφίζουμε υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική D υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 και 60 στη συνέχεια, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 62 της κυρίας Βιλπάου, υπέρ, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68 στη συνέχεια. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να κάνουμε μια παλήθευση όμως γιατί δεν είμαι σίγουρος από πλευρά σοσιαλιστών τι γίνεται. Για την 68 άρχεται η ψηφοφορία, ψήφισαν όλοι, πέρασε τη ψηφοφορία, εγκρίνεται. Συμβιβαστική F, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία G υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 77 με προφορική τροπολογία του κυρίου Κοχ. Την έχετε. Υπάρχει κάποια ένσταση για την προφορική τροπολογία. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέτζι 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται, 82 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 83 υπέρ, κατά, αποχές. Να κάνουμε μια παλήθευση για την 83, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 84 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ρέτζι 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 85 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ρέτζι 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ρέτζι 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ρέτζι 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ρέτζι 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 86 υπέρ,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 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. 35 ψήφοι υπέρ, 2 κατά και 1 αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν. Συγχαρητήρια κύριε Κράμερ. Περνάμε τώρα στην γνωμοδότηση του κυρίου κουσιέρη, Τροποποίηση της οδηγίας 92 του 2011 σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Ξεκινάμε με την 21 από τον κύριο Κράμερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πολύ καλά τα Πάσκρα, ε, Μάικολ. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. 2 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να κάνουμε μια επαλήθευση για την 23 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 24-25 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 26 της κυρίας Βουίλς υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση για την 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να κάνουμε και γι' αυτό έναν έλεγχο. Νομίζω την ίδια πλειοψηφία έχουμε, αλλά να κάνουμε έναν έλεγχο γιατί... Ψήφισαν όλοι, πέρας της ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 3. του εισηγητή, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 29 και 4 που είναι πανομοιότυπες υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Κατά τμήματα 30 τώρα, όλο το κείμενο χωρίς τη φράση The Social Impact End και μετά το δεύτερο τμήμα είναι το The Social Impact End. Το τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να κάνουμε έναν έλεγχο, αλλά νομίζω ότι απορρίπτεται. Έχει νόημα το δεύτερο τμήμα. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται, επομένως, το δεύτερο τμήμα δεν έχει νόημα. 31 και 32 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να κάνουμε μια παλήθευση για την 5 του συντάκτη υπέρ. Ε, συγγνώμη, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 6 του συντάκτη υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται, 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 34 υπέρ, κατά, αποχές, να κάνουμε μια επαλήθευση για τη 34, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 37. Αυτά τα περιβόητα με και σάλ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά αποχές. Να κάνουμε μια παλήθευση για την 7, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 40-41 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 8 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνονται, εγκρίνεται, 42 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος για τη 42, νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά άρχεται η ψηφοφορία παρόλα αυτά. Ψήφισαν όλοι, πέρασε της ψηφοφορίας, απορρίπτεται όντως, 43 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 45 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 46 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθεση για τη 46, άρχεται η ψηφοφορία, ψήφισαν όλοι, πέρασε της ψηφοφορίας, απορρίπτεται, 48, 50 ε, και 51 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέραση η ψηφοφορίας, απορρίπτεται, 47, 49 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος και για αυτές, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτονται λόγω ισοψηφίας. 51-52 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική α. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται.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 να κάνουμε μια επαλήθευση για την 63, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 64 υπέρ. 64 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επαλήθευση. Δεν είμαι πολύ βέβαιος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος για την 67 παρακαλώ, εγκρίνεται νομίζω. Να δούμε όμως τι γίνεται στο ΕΛΚ, ψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Υπέρ 68, κατά, Αποχές ε, απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παραρτήματα 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να κάνουμε μια παλήθευση για την 71. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 74, 75 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 11 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 και 17 καταπίπτουν. 20 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα η τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 34 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Κουσχέρη. You have the hearing now. Now move on to the hearing. If we just... Θα περάσουμε τώρα στην ακρόαση. Δώστε μας μόνο ένα λεπτό και δίνουμε και σας ένα λεπτό για να βρείτε τη θέση σας.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 Okay, colleagues, Λοιπόν, συνάδελφοι, να μην καθυστερήσουμε. Θα είναι καλό για όλους μας. Περνάμε λοιπόν στην μίνι ακρόαση για τις ε, νέες μορφές ε, καθαρής ενέργειας για τις μεταφορές. Θα δώσουμε πρώτα το λόγο στον κύριο Νίδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα ακούσουμε παρουσιάσεις τον κύριο Κρίστη, την πλατφόρμα για τον εξελικτρισμό των ηχεσίων μεταφορών, του κυρίου Μάτζ, αν το λέω σωστά, NGVA Europe και από τον κύριο Ζιόλεκ από την HYER, κύριος Ρίκο από την Black Alliance και ο κύριος από την Ένωση Κατασκευαστών ε, Αυτοκινήτων. Αυτό είναι το πρώτο πάνελ. Θα έχουμε μετά ένα γύρο ερωτήσεων-απαντήσεων και στη συνέχεια περνάμε στο δεύτερο πάνελ από τον κύριο Λάρος, κύριο Μπίλιετ, από το IRU, κύριος Γκουίντα από την Ένωση ε, Δημόσιων Μεταφορών, UITP, κύριος Χάουν από τις Ευρωπαϊκές Πόλεις και Περιφέρειες και κύριος Μάρτενς, αυτός που έχει τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ξεκινάμε λοιπόν με τον κύριο Ολιβιέ Ονίδη από πλευράς Επιτροπής. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Να πω εξ αρχή ε, σε όλους τους ομιλητές ότι στις ακροάσεις ε, είμαι πάρα πολύ αυστηρό με το χρονοδιάγραμμα. Επομένως, ε, μείνετε στο χρόνο που έχετε, αλλιώς θα σας κόβω το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Έχω συνηθίσει την αυστηρότητά σας, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω εδώ, μέσα σε αυτή τη μήνυα ακρόαση που είναι, έχει θέμα εξαιρετικά σημαντικό για μας Βεβαίω είμαστε εδώ κυρίω για να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονε, επομένω θα είμαι σύντομο, Μερικές παρατηρήσεις μόνο από πλευρά μας. Η πρόταση που έχετε εδώ για την καθαρή ενέργεια για τι μεταφορές είναι πρώτα απ' όλα μια ε, δυνατότητα, μια ευκαιρία για να δώσουμε στον τομέα των μεταφορών την ευκαιρία να ξεφύγει από την μία και μοναδική πηγή εφοδιασμού, δηλαδή το πετρέλαιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο κινούμε ε, σε πολλά επίπεδα. Είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια του εφοδιασμού και ενέργειας ε, και στο πλαίσιο της ευρύτερης ατζέντας μας για το περιβάλλον και για την κλιματική αλλαγή. Αλλά πιο σημαντικό από όλα είναι ότι είναι πολύ σημαντικό για την ε, οικονομία μας. Γιατί δαπανούμε ένα δις την ημέρα για την εισαγωγή πετρελαίου. Πάνω το 50% πηγαίνει στον τομέα των μεταφορών είναι θεμελιώδη σημασία για την ανταγωνιστικότητα τη βιομηχανία μα, δηλαδή η ανάπτυξη ε, εναλλακτικών πηγών ενέργεια και καυσίμων. Ε, είμαστε βέβαια επικεφαλής ε, στον αγώνα για την ανάπτυξη τέτοιων μορφών ενέργειας, αλλά ο ανταγωνισμός είναι πολύ δύσκολος και από πέρυσι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια νέα αγορά με επιπλέον φορείς. Και τέλος είναι εξαιρετικά θετικό και για τους χρήστες, για τον κόσμο. Γιατί με αυτές τις νέες ε, μορφές οχημάτων έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να αλλάξουμε τις ε, συνήθειές μας και τον τρόπο που κινούμαστε για να ακολουθήσουμε μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση. Τρεις είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις κατά τη γνώμη μας. Πρώτον, ε, να αφορά αυτή η προσπάθεια όλα τα καύσιμα όχι να έχουμε δηλαδή μόνο μια νησίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαφόρων ε, τεχνολογιών που τελικά δεν ε, θα είναι συμβατέ μεταξύ του. Να καλύπτονται λοιπόν όλα τα καύσιμα και όλες ε, οι μορφές μεταφορών. Γι' αυτό και η πρόταση πράγματι καλύπτει όλες τις μορφές από τα βιοκαύσιμα ε, στην, ε, στις αερομεταφορές μέχρι το υγροποιημένο στις ε, θαλάσσιες μεταφορές. Χρειαζόμαστε δεύτερον και μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση. Δεν θέλουμε δηλαδή τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν διαφορετικές τεχνολογικές λύσεις και ούτε θέλουμε την διάδοση μη συμβατών μεταξύ τους προτύπων. Χρειαζόμαστε σε μια, μια αγορά στο μέγεθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γι' αυτό και προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να επιβάλλουμε κοινά πρότυπα με τους κατάλληλους μηχανισμούς και βασιζόμαστε και στο συντονισμό εθνικών σχεδίων για την ανάπτυξη αυτών των εναλλακτικών καυσίμων. Τρίτο, χρειαζόμαστε πολύ συγκεκριμένους στόχους. Το βασικότερο ε, στοιχείο σήμερα είναι η ανάπτυξη υποδομών για την ε, φόρτιση ή τον ανεφοδιασμό ε, καυσίμου και αυτό είναι απαραίτητο για τους ε, επενδυτές. Δηλαδή το να υπάρχει ένα δεσμευτικό πλαίσιο το οποίο αποτελείται από πολύ συγκεκριμένους στόχους τουλάχιστον μέχρι το 2020. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Νονίδη. Να περάσουμε τώρα στους εμπειρογνώμονες. Πρώτος που θα πάρει το λόγο είναι ο κύριος Edward Christie επικεφαλής ε, οικονομολόγος ε, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Σιδηροδρόμων ε, και εκ μέρους της πλατφόρμας για τον εξελεκτρισμό των χερσών μεταφορών. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα σε ό,τι αφορά την πλατφόρμα για τον εξελεκτρισμό χερσαίων μεταφορών. Ε, είμαστε, ε, ασχολούμαστε με ολόκληρο το τομέα αυτής της βιομηχανίας ε, μαζί με τις τοπικές αρχές. Θέλουμε να προωθήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση με ένα εξελεκτρισμένο διατροπικό σύστημα μεταφορών. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Και αυτό είναι και το μέλλον του ευρωπαϊκού συστήματος υπηρεσιών μεταφορών. Να σας δείξω πρώτα δύο γραφήματα που δείχνουν ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικός ο εξελεκτρισμός. Βλέπετε εδώ τις περιβαλλοντικές επιδόσεις. Η Διεθνής Ένωση Ενέργειας το 2011 μας έχει δώσει αυτά τα στοιχεία. Είχε εκπονήσει έκθεση για τις μελλοντικές προοπτικές του φυσικού αερίου. Και εδώ βλέπετε αυτό ε, που, αποκαλούμε εκπομπές well to wheel, από το φρέαρ ε, στη, στα οχήματα. Για να δείτε πόσο ακριβώς ε, έχουν οι επιδόσεις σε επιμέρους περιφέρειες. Αν, δι, αν είστε στις ΗΠΑ ή στην Κίνα ή στην Ινδία, έχετε ένα ενεργειακό μείγμα που είναι πολύ πιο έντονο σε φορά τις εκπομπές σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά. Επομένως, εκεί είναι λιγότερο ελκυστική ηλεκτρι... ελκυστικός ο Όμως, σε μια αγορά όπως την Ευρώπη, ο εξελεκτρισμός ε, δίνει τεράστια ωφέλη σε ό,τι αφορά τι εκπομπές. Οποιαδήποτε άλλη, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική, όπως βλέπετε εδώ και με το βέλος. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο επιχείρημα για ε, τις ηλεκτρικές μεταφορές. Μετά, σε ό,τι αφορά την εξάρτηση, προφανώς και η ε, ασφάλεια στην ενέργεια ε, δεν αφορά μόνο την, ε, την εξάρτηση αλλά και την εξέβρεση των καυσίμων. Γι' αυτό και συμφωνούμε με την προσέγγιση της Επιτροπής να εξετάσουμε πολλά και διαφορετικά καύσιμα, όχι δηλαδή να επικεντρωθούμε σε ένα μόνο. Όμως να έχουμε κατά νου ότι και πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ίδια με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τουλάχιστον προς το παρόν δεν έχουμε αυτή την έκρηξη στον τομέα του συστολιθικού αερίου που θα μας δώσει νέες δυνατότητες. Γιατί αν δείτε, ε, την εξάρτηση, η εξάρτηση των ΗΠΑ για πετρέλαιο και φυσικό αέριο μειώνεται και γίνεται μάλιστα και χώρα εξαγωγός ε, φυσικού αερίου, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την αντίθετη τάση αύξηση τη εξάρτηση. Και κοντεύουμε να φτάσουμε στα ίδια επίπεδα εξάρτηση για το φυσικό αέριο με το πετρέλαιο. Επομένω, το να αλλάξουμε ε, από το πετρέλαιο στο φυσικό αέριο δεν θα γίνουμε λιγότερο εξαρτημένοι. Δεν θα μειωθεί λοιπόν το πρόβλημα τη εξάρτησή μα. Αυτά τα δύο στοιχεία πρέπει να τα έχουμε κατά νου μαζί και με άλλα βεβαίω. Όμω είναι σημαντικά επιχειρήματα για την στροφή προς ε, τι ηλεκτρικέ μεταφορέ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόταση τη Επιτροπής, ε, τη χαιρετίζουμε. Ε, είναι μια καλή πρωτοβουλία από πολλέ επιτυχές. Είναι αρκετά ευρεία, καλύπτεται και η ναυτιλία. Όμως, καθώς η δική μας πλατφόρμα είναι πολυτροπική, ε, θεωρούμε ότι μπορούν να γίνουν περαιτέρω βήματα. Θέλουμε λοιπόν να προσθέσουμε κάποια στοιχεία στην πρόταση. Θα προτείνουμε λοιπόν ε, τροπολογίες ε, για να προσθέσουμε νέες διατάξεις που θα λαμβάνουν υπόψη αυτή την πολυτροπική διάσταση σε ό,τι αφορά τη σύνδεση των νέων υποδομών με τις δημόσιες μεταφορές και τους υδροδρόμους και τη σύνδεση με τα δίκτροχα οχήματα. Ε, άλλη διάσταση είναι στη συμμετοχή στην πλατφόρμα μας. Έχουμε και ε, παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Γι' αυτό εξετάζουμε ιδιαίτερα τις διατάξεις στο άρθρο 4 για την ε, παροχή, την μέτρηση, την ευφυή μετρήση και το καθεξής. Θα έχουμε λοιπόν κάποιες ε, προτάσεις από αυτού. Θα έχουμε και για τους ε, υποχρεωτικούς ε, στόχους, αλλά γενικά συμφωνούμε. Για τα σημεία ανεφοδιασμού πεπιασμένου φυσικού αερίου θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να αφορά τα κράτη-μέλη και να μην υπάρχουν ευρωπαϊ... υποχρεωτικοί περιορισμοί σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και συμφωνούμε και τη γενική κατεύθυνση εναρμόνιση των τεχνικών προτύπων για τον ανεφοδιασμό ή τη φόρτιση. Τώρα, λίγο πιο συγκεκριμένα και εν συντομία. Θέλουμε να έχουμε διατάξεις φιλικές προς τις επιχειρήσεις ε, για τον εφοδιασμό ενέργειας ε, και τη φόρτιση με κατάλληλη ενημέρωση είναι πολύ σημαντικό ε, ναι, να υπάρχει διαφανής ενημέρωση και των καταναλωτών ε, και σε ό,τι αφορά τις τιμές και να έχουμε μια δυνατότητα ε, επικοινωνίας δύο κατευθύνσεων μεταξύ των οχημάτων και του δικτύου. Τέλο, εναρμόνιση των τεχνικών προτύπων για την εφόρτιση. Συμφωνούμε με την πρόταση Επιτροπή να επικεντρωθούμε στι μορφέ τύπου 2 για το fast charging δεν θέλουμε να δοθεί έμφαση μόνο στο πρότυπο Combo 2 ε, και δεν πρέπει να αποκλειστεί και το υπάρχον ε, πρότυπο καντίμου. Ευχαριστώ. Much, Ευχαριστούμε τον κύριο Κρίστη. Ο κύριος Μάτζ. Από ε, την NGVA Europe. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ε, έντιμα και εξέχοντα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με μεγάλη χαρά σας παρουσιάζω τις προτάσεις μου. Δεν πρόκειται να σας πω τι τροπολογίες πρέπει να ψηφίσετε και τι όχι. Απλώς θέλω να σας πείσω να μας υποστηρίξω και να σας, εξηγήσω, να σας γιατί το μεθάνιο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στις μεταφορές. Εκπροσωπεί μια οργάνωση που προωθεί τα περιβαλλοντικά φιλικά ε, καύσιμα η μοριακή δομή του μεθανίου που είναι άνθρακα υδρογόνο 4 ε, παίζει σημαντικό ρόλο επειδή έχει χαμηλότερο ποσοστό άνθρακα στο να μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Επίσης μειώνεται και ο θόρυβος από, τα, ε, από τους κινητήρες που χρησιμοποιούν μεθάνιο και λειτουργεί σε κάθε είδους ε, μορφές οχημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντικό το θέμα των ε, εκπομπών και μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε και τη χρήση βιομεθανίου. Λοιπόν, μπορούμε να έχουμε κανονικό μεθάνιο ή μεθάνιο σε υγροποιημένη μορφή. Δεν έχουμε κανένα λόγο να έχουμε επενδύσεις για να μετατρέψουμε τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν για υγροποίηση και αυτό το τμήμα της πρότασής μας. Επιπλέον, μπορείτε να παραγάγεται συνθετικό φυσικό αέριο με την τεχνολογία αυτή από, για τη χρήση ηλεκτρισμού από, για, από ανανεώσιμες, πηγές που δεν μπορούμε να τις ε, αποθηκεύσουμε την πρόσθετο ηλεκτρισμό. Χρησιμοποιείται λοιπόν τον ε, ηλεκτρισμό για παραγωγή υδρογόνου που μετά οδηγεί σε παραγωγή μεθαρίου το οποίο μπορεί να διανυμηθεί και να χρησιμοποιηθεί στις μεταφορές. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν το θέμα των εκπομπών. Και βλέπετε εδώ ότι τα οχήματα με φυσικό αέριο μπορούν να είναι εξίσου καθαρά όσο τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αν λάβουμε και την παραγωγή, υπόψη και την παραγωγή από ανανεώσιμες ενέργειες. Επίσης λοιπόν θεωρούμε ότι μπορούμε να τροποποιήσουμε και τη συμμετοχή τους στις ανανεώσιμες ενέργειες. Είναι σημαντική και η ποιότητα της ατμόσφαιρας. Ζούμε όλοι εδώ πέρα σε αυτό το μαύρο κομμάτι της Ευρώπης που βλέπετε εδώ και καταλαβαίνετε περισσότερο γιατί. Αλλά η χρήση ε, του υποπίεση φυσικού αερίου στις πόλεις, ιδίως στα δημόσια οχήματα, στα σκουπιδιάρκα κτλ. μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ να μειώσουμε την ε, ρήπανση. Χρειαζόμαστε αυτή την ε, υποδομή γιατί θα έχουμε και τη μισή, το μισό επίπεδο θορύβου σε σχέση με τη χρήση του ντίζελ. Φυσικά είναι και ένα θέμα που έχει να κάνει με τις τιμές των καυσίμων. Ο καταναλωτής βασίζεται σε ένα οικονομικό μοντέλο οι τιμές των, ε, το ψαλίδα μεταξύ πετρελαίου και φυσικού αερίου αυξάνεται. Ίσως επειδή υπάρχει το αέριο από σχιστολή του στις Ηνωμένες Πολιτείες θα αλλάξει αυτή η αγορά. Οι υποδομές όπως ξέρετε έχουμε τους αγωγούς αυτούς που διασχίζουν όλη την Ευρώπη. Υπάρχει υποδομή για ενεργειακούς θερματικούς σταθμούς έχουμε όλο και περισσότερη διαθεσιμότητα υγροποιημένου φυσικού αέριου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Ρήνο και τον ε, Δούναβη για να κυκνούνται με μαούνες στους εσωτερικούς υδάτινους δρόμους. Μπορούμε έτσι να φτιάξουμε διαδρόμους για μεταφορά ενέργεια στην Ευρώπη που είναι πιο αποτελεσματική από τους σιδηρόδρομους και τα φορτηγά. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι υποδομές στην Ευρώπη. Όλες οι χώρες της Ευρώπης ακόμα έχουν υποποίηση φυσικό αέριο είναι κατακαιρματισμένη η κατάσταση, γι' αυτό χρειάζεται να εναρμονίσουμε καλύτερα την αγορά. Μόνο 0,5% είναι το ποσοστό της αγοράς, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να φτάσουμε στο 5% το 2020. Έχουμε μονάχα περιορισμένο αριθμό οχημάτων, είναι πολύ δύσκολο να το δει κανείς. Έχουμε 700.000 στην Ιταλία, 100.000 στη Γερμανία, 9.900 σταθμούς. Δύο τρίτα της αγοράς λοιπόν σε σταθμούς ε, φυσικού αερίου είναι εκεί. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι περισσότερη υποδομή. Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ε, πιστεί ότι η χρήση του φυσικού αερίου είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μειωθούν και οι εκπομπές. Βλέπετε αυτοκίνητα όπως το Volkswagen αυτό, το οποίο θεωρήθηκε αυτοκίνητο της ε, χρονιάς. Το Fiat κέρδισε με το πιο πράσινο αυτοκίνητο της χρονιάς εδώ μειώνουμε την ε, αποτελεσματικότητα των οχημάτων αυτών γιατί έχουν και μηχανή εφεδρική βενζινοκινητήρα. Εάν έχουμε μονάχα <clears throat> το φυσικό αέριο όμως θα μειώσουμε πάρα πολύ σημαντικά τις εκπομπές φυσικού ε, αερίων του θερμοκηπίου. Η Ευρώπη παίζει πρωταρχικό ρόλο, είναι ηγέτη σε παγκόσμιο επίπεδο οι εταιρείε μα είναι λοιπόν ηγέτε στην αυτοκινητοβιομηχανία. Σημαντική πληροφορία και για του καταναλωτέ. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ότι το φυσικό αέριο είναι το πιο το πεπιεσμένο, το πιο ε, φτηνό. Όταν μιλάμε λοιπόν για, το πεπιασμένο φυσικό αέριο, δεν είναι μονάχα κάτι το οποίο μα ενδιαφέρει στα αυτοκίνητα, χρειαζόμαστε και υγροποιημένο αέριο για τα μεγάλα οχήματα, δεν δηλαδή είναι θέμα ενεργειακή. Ε, ε, ενέργεια συνολική, αλλά ενεργειακή πυκνότητας. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε και το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Έχετε σταθεί παρόντες τον προηγούμενο Μάιο για το σχέδιο των διαδρόμων για το φυσικό αέριο και ξέρετε τη σημασία. Το στόχος του να υπάρχει να υπάρχουν διαφορές ε, αποστάσεις 400 χιλιόμετρων και αντίστοιχα 150 για το πεπιεσμένο αέριο είναι ο στόχος μας. Και κλείνω κύριε Πρόεδρε, αυτοί είναι οι στόχοι που πρέπει να υποστηριχτούν. Πρέπει να θυμόσαστε ότι το πεπιεσμένο φυσικό αέριο συνδέεται με ένα αγωγό και το υγροποιημένο με κρυογενικές εγκαταστάσεις. Είναι πάντως σημαντικές εγκαταστάσεις. Άμα δούμε τις διάφορες λύσεις για τις μορφές αυτές φυσικού αερίου, είναι πάρα πολύ σημαντική η διατροπικότητα. Είναι σημαντικό να μπορούμε να έχουμε <clears throat> ε, σταθμούς επαναφόρτησης και το μεθάνιο μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Τα προϊόντα αυτά είναι διαθέσιμα σε ανταγωνιστικές τιμές. Είδατε λοιπόν τη διαφορά στα αυτοκίνητα, έχουμε σημαντικές τεχνολογίες, είναι μια αγορά που αναπτύσσεται, νομίζουμε ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε το 20% στο 2050, πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη υποδομή. Τέλος, υποστηρίξτε λοιπόν το πακέτο για την καθαρή ενέργεια στις μεταφορές ήταν το αποτέλεσμα προσπαθειών πολλών ετών όπου η Κομισιόν συνεργάστηκε με εμπλεκόμενους όπως είναι ο δικός μου φορέας και η πρωτοβουλία αυτή είναι πολύ σημαντική και κρατήστε την ε, το χρονοδιάγραμμα. Θα πρέπει ήδη να είχε εγκριθεί αυτό. Πρέπει να προωθήσουμε λοιπόν αυτά τα καύσιμα και θα πρέπει να προωθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζιόλεξ στη συνέχεια, ο οποίος είναι πρόεδρος ε, της ε, HYER για τη χρήση του υδρογόνου. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι καλημέρα. Θα προσπαθήσω να μιλήσω όσο γρήγορα και ο προηγούμενος Για την Χάιερ λοιπόν να σας πω δύο λόγια. Εδώ έχετε ένα χάρτη με όλα μας τα μέλη. Εκπροσωπούμε 40 περιφέρειες ανά την Ευρώπη που ασχολούνται με θέματα χρήσης υδρογόνου. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω όλα τα στοιχεία εδώ. Όλες αυτές οι περιφέρειες συνεργάζονται για την ηλεκτρική κινητικότητα αλλά για διαφορετικούς λόγους η καθεμία και αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε όλα τα μέλη μας ζητούν να εργαστούμε σε αυτά τα τρία βασικά σημεία δράσης. Καταρχάς, να διευκολύνουμε συστάσεις πολιτικής που βασίζονται σε αυτά στοιχεία, να αναπτύξουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο υποστήριξης και να έχουμε μια εύρωστη ε, αγορά. Να σας πω δύο λόγια τώρα για τις γενικές θέσεις της Higher για την ε, πρωτοβουλία για την καθαρή ενέργεια. Καταρχάς, ε, να σας πω ότι τα, μέλη της Higher ε, συμμερίζονται και φυσικά υποστηρίζουν τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει και να επιταχύνει την εφαρμογή της ε, χρήσης κυψελών ε, ε, καυσίμου υδρογόνου και τη ηλεκτρικής κινητικότητας και θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Συμφωνούμε ότι η προτυποποίηση είναι βασικό θέμα για να καλύψουμε κάποιες από τις βασικές προκλήσεις, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος, για να επιταχύνουμε τις υποδομές, ε, τη βελτίωση των υποδομών και να κινητοποιήσουμε τις οικονομίες κλίμακες ε, και να μειωθεί το κόστος φυσικά έχουμε διαπιστώσει σε αρκετά προγράμματα ότι οι διαφορετικές προδιαγραφές είναι ε, μία από τις μεγαλύτερες ε, προκλήσεις και αποτελούν πρόσκομα στην ε, εντατικότερη συνεργασία και αυτό φάνηκε σαφέστατα σε ένα-δυο προγράμματα που κάναμε. Να σας πω κάποια πράγματα για τις δεσμεύσει μας, για τους στόχους, για, τις, ε, ε, για την καθαρή ενέργεια. Θεωρούμε ότι οι στόχοι μπορεί να είναι επιτυχείς μόνο αν οι δεσμεύσει γίνονται αποδεκτές από όλους τους ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων και των διαχειριστών των συστημάτων μεταφοράς και ενέργειας. Είναι πάρα πολύ συμμετοχή σημαντική συμμετοχή και προσπαθούμε να την ενισχύσουμε όπου είναι δυνατόν. Επίσης, οι φιλοδοξίες και οι στόχοι θα πρέπει να αναγνωρίζουν και ε, τους τοπικούς και περιφερειακούς ε, στόχους ε, και τις συνθήκες που επικρατούν και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να δώσουμε και αυτή τη διάσταση. Οι στόχοι πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία και σε εμπειρίες ή δυνατόν σε συγκεκριμένα έργα και προγράμματα και εδώ θα θέλαμε να συνεισφέρουμε και εμείς με ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που έχουμε συστήσει με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ηλεκτρικής Κινητικότητας. Αυτό σχετίζεται με το στόχο υπαριθμών 3 να έχουμε ε, συγκεκριμένα εύρωστα ε, στοιχεία διανομής ε, της αγοράς. Ε, αυτό έχει γίνει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει συσταθεί το 2012 και είναι ένα ε, στοιχείο το οποίο διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και συντονισμένες δράσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε λοιπόν ε, τι μας παρακινεί και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και τι διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από αυτές τις πρακτικές. Προσπαθούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους διάβλους για να έχουμε συγκεκριμένη κάλυψη ε, και να γίνει αυτό ένα βασικό εργαλείο για όσους χαράσουν πολιτική σε όλα τα επίπεδα, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν το σχεδιασμό των υποδομών, να αναλύουν τα δεδομένα και να κάνουν συστάσεις. Να σας καλέσω επίσης ε, στο τελευταίο μας, ε, στο επόμενο εργαστήριό μας που θα γίνει εδώ στις ε, Βρυξέλλες στις 24 Ιουνίου. Τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό, κάποιες συστάσεις που βασίζονται στα πρώτα αποτελέσματα της ε, μελέτης του παρατηρητηρίου. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι προκειμένου να υποστηρίξουμε όσους χαράσουν πολιτική για να καθορίσουν τις ε, σημαντικές ε, στρατηγικές για να προχωρήσει η υποδομή, θα πρέπει να βρούμε τις τάσεις, ε, να εξετάσουμε διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα και να υποστηρίξουμε συγκεκριμένα προγράμματα, διότι όπως σας είπα είναι πολύ διαφορετικά τα στοιχεία ανά την Ευρώπη. Ο καθένας θέλει να περάσει την ηλεκτροκίνηση για τους δικούς του λόγους και εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε την οδηγία όσο το δυνατόν περισσότερο. Επίσης ε, πρέπει να δούμε επίσης ε, πώς μπορεί να γίνεται επαναφόρτιση και χρήση ε, των καυσίμων. Ε, θεωρούμε επίσης ε, πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώς έχει το τοπίο. Είναι πολύ διαφορετικό να έχουμε μια περιοχή της υπαίθρου ή μια αστική περιοχή με διαφορετικό κλίμα. Δεν μπορούμε να έχουμε μια ενιαία προσέγγιση για όλα. Πρέπει να γνωρίζουμε τι χρειάζεται ο κάθε πελάτης και τι κάνει. Και επίσης είναι πολύ σημαντικές οι σχέσεις μεταξύ των περιφερειακών και εθνικών αρχών μεταφορών και ενέργειας για να μπορούν να καθορίσουν και κάποιους κοινούς παρανομαστές. Ε, χρειαζόμαστε επίσης κατευθυντήριες γραμμές και καθοδήγηση για να έχουμε εναρμονισμένη πρόωθηση των υποδομών και ε, χρειάζονται φυσικά και χρηματοδότηση από αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα. Να σας ε, πω λοιπόν ότι εμείς ε, υποστηρίζουμε πλήρως την οδηγία, η Χάιερ είναι διατεθειμένη να βοηθήσει και ελπίζουμε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ζιόλεξ. Στη συνέχεια ο κύριος Κλοντρικό από το EV Plug Alliance. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η EV Plug Alliance είναι μια ένωση ε, επιχειρήσεων για την προώθηση ασφαλούς, ε, διαλειτουργικής ε, και λύσεων που έχουν, είναι αποτελεσματικές και ως προς το κόστος για καθαρές μεταφορές. Ε, οι υποδομές επαναφόρτηση είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι περισσότερες υπάρχουν. Υπάρχουν ε, ε, εργοστάσια, δίκτυα διανομής που διανέμουν ηλεκτρική ενέργεια σε κτίρια και σε επιχειρήσεις και φυσικά αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται εκ νέου νέα υποδομή. Αυτό το οποίο δεν διαθέτουμε είναι σημεία επαναφόρτισης. Σημεία τα οποία θα επιτρέπουν ε, σε ένα αυτοκίνητο να χρησιμοποιεί το δίκτυο διανομής και να ε, κάνει επαναφόρτιση με ασφάλεια. Αυτό ακριβώς εννοούμε λοιπόν εμείς, ε, να υπάρχουν διάφορα σημεία επαναφόρτισης τα οποία θα επιτρέπουν στον καθένα να κάνει επαναφόρτιση είτε αργή είτε ταχύ επαναφόρτιση στο μέλλον. Εκτιμάται ότι το 90% αυτών των σημείων επαναφόρτισης θα βρίσκονται σε σπίτια και σε κτίρια και ένα 10% μόνο θα βρίσκονται σε δημόσιους χώρους, ε, σε χώρους στάθμευσης ή σε χώρους επαναφόρτισης. Και η ενσωμάτωση αυτών των σημείων παραφόρτισης σε κτίρια και σε ε, κατοικίες είναι η βασική απέτηση. Οι υποδομές αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές για να επιταχύνουμε την έγκριση της ηλεκτρικής κινητικότητας. και αυτό ακριβώς και καλωσορίζουμε το στόχο της οδηγίας να επιταχύνουμε την ε, ε, χρήση ενός ε, μεγάλου διαλειτουργικού εφιούς ε, δικτύου υποδομών επαναφόρτησης, το οποίο είναι σημαντικό για την ηλεκτρική κινητικότητα και είναι αυτό το οποίο μας λείπει αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η οδηγία αυτή να ολοκληρωθεί ταχύτατα και να εφαρμοστεί και η, εφαρμοστή, και η εφαρμογή της να είναι εύκολη για όλες τις χώρες. Θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία μπορούμε να επιφέρουμε κάποιες βελτιώσεις ε, στην οδηγία, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις ε, κατά την έγκρισή της. Η EV Plug Alliance θέλει να συνεισφέρει στην συνένεση και στην επιτάχυνση της έγκρισης της οδηγίας. Τι έχουμε κατά νου. Η οδηγία επέλεξε μια τεχνολογία, τη λεγόμενη τύπου 2, για την διαλειτουργικότητα, για τις ε, ε, συνδέσεις υποδομών. Τώρα, το να το εγκρίνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μια οδηγία που θα είναι συμβατή με τις ε, πρακτικές ασφαλείας ε, της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και προκειμένου να επιτευχθεί αυτό υπάρχει μια πολύ απλή λύση. Η οδηγία θα πρέπει να περιγράφει τη χρήση και της βασικής χρήσης πρίζας τύπου 2 και επίσης ε, κάποια ε, στοιχεία διακοπής ασφαλείας ε, τα οποία χρειάζονται σε κάποιες χώρες. Και όλα αυτά θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατά φυσικά με τις μπρίζες τύπου 2 που διατίθεται αυτή τη στιγμή. Ο κλάδος λοιπόν είναι διατεθειμένος να βοηθήσει για την ταχεία βιομηχανοποίηση με αποδοτικός προς το κόστος τρόπο και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προβολή και να διασφαλίσουμε ότι θα συμπεριληφθεί το στοιχείο αυτό στην οδηγία. Αυτό που έχει σημασία είναι η λύση αυτή να ανταποκρίνεται στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπάρχει μια ενιαία πρίζα επαναφόρτησης, ε, ώστε να μπορεί κάποιος να επαναφορτήσει το όχημά του οπουδήποτε στην Ευρώπη. Υπάρχουν βέβαια και κάποια σημεία τα οποία χρήνουν διευκρίνησης και θα πρέπει ίσως να προσέξουμε λίγο περισσότερο στην οδηγία. Το πρώτο είναι ότι υπάρχουν κάποιοι επενδυτές οι οποίοι επένδυσαν ε, εκ των προτέρων και ενδιαφέρονται για αυτή την ηλεκτρική κινητικότητα και δεν θα πρέπει να τιμωρήσουμε αυτούς τους ε, ε, πρώτους χρήστες από την, με την νέα οδηγία. Η υποχρέωση λοιπόν ε, της ε, αλλαγής ε, των υφιστάμενων υποδομών πρέπει να είναι περιορισμένη απλώς και μόνο στις δημόσιες υπονομές και δεν θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση να γίνεται αυτό στον ιδιωτικό χώρο εάν υπάρχουν άλλες δυνατότητες και εμεί θεωρούμε ότι υπάρχουν άλλες δυνατότητες και πρέπει να δοθεί και επαρκής χρόνος να προσαρμοστεί κάποιος στις αλλαγές ε, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του και το χρονοδιάγραμμα που έχει καθορίσει η αυτοκινητοβιομηχανία για τη μετατροπή ε, των στιγμίων επαναφόρτησης. Γι' αυτό ακριβώς προτιμούμε τον ε, τρόπο 3 που είναι ένας τρόπος εφιούς επαναφόρτησης που θα μας επιτρέψει να έχουμε και προηγμένη διαχείριση ενέργειας. Η δυνατότητα όμως επαναφόρτησης ε, με τον τρόπο 1 και τρόπο 2 που είναι ήδη ενισχύ θα βοηθήσει να καθησυχάσουμε τους χρήστες κυρίως τα πρώτα χρόνια χρήσης της νέας υποδομής ε, διότι θα είναι περιορισμένη η χρήση και είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κάποιος να κάνει επαναφόρτωση σε διάφορα σημεία. Επίσης θα είναι πολύ χρήσιμο για ελαφρά οχήματα όπως για παράδειγμα δίκυκλα. Η οδηγία λοιπόν δεν θα πρέπει να αποκλείσει και το ενδεχόμενο να κάνει κάποιος επαναφόρτηση με τον τρόπο 1 ή 2 για να μπορούν να ε, εξυπηρετηθούν και οι χρήστες. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταίος ομιλητής ο κύριος Πέτρε Ντελόεση εκ μέρους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Κατασκευαστών Αυτοκινήτων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Όπως Αναφέρθηκε εκπροσωπώ την ΑΣΕΑ που εκπροσωπεί όλους τους ε, και τους 16 μεγάλους ε, κατασκευαστές στην Ευρώπη. Βασικό μας ε, μότο είναι ότι όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα στην κατασκευή και αυτό θα είναι εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο κατά την εξέταση των στοιχείων της Λοιπόν, για τα αναλλακτικά κάψιμα βλέπουμε ότι στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής ε, για αυτά τα οχήματα καθαρή ενέργεια σημαίνει ότι επικεντρωνόμαστε ε, στην βελτίωση των ε, μηχανών καύσης αλλά και στα αναλλακτικά καύσιμα και θεωρούμε ότι οι μεταφορές θα χρειαστούν διαφορετικές τεχνολογίες και ένα πολυτροπικό σύστημα. Είναι καλό λοιπόν που δεν επικεντρωνόμαστε μόνο σε μία μορφή ενέργειας. Η αρχή της ε, ενεργειακής ουδετερότητας είναι σωστή, πρέπει να διατηρηθεί και ωφελεί και εμάς και τους πελάτες μας. Γιατί τελικά ο καταναλωτής είναι αυτός που θα αποφασίσει τι θα αγοράσει, αν θα είναι ένα ε, σύνηθες ε, όχημα ή ένα ηλεκτρονικό ας πούμε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις, το σιδηρόδρομο εναλλακτική ενέργειας, αυτό είναι ένα ζήτημα μακροχρόνιας πολιτικής, απαιτείται συντονισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ε, διαφόρων εθνικών στρατηγικών. Χρειάζεται θέσπιση η τυποποίηση σε όλη την Ευρώπη και υποδομές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι η επιτυχής μετάβαση προς ε, αυτή την ηλεκτρική κίνηση δεν αφορά μόνο τους κατασκευαστές αλλά όλους τους κλάδους. Εμείς βεβαίως ε, εκφράζουμε τη δέσμευση να ε, συμβάλλουμε, όμως πρέπει να βελτιωθούν τα οχήματά μας και σε τέτοιου σιδηροδρόμου εναλλακτική ενέργεια για να ικανοποιούνται και τα αιτήματα των καταναλωτών. Όμω Πράγματι πρέπει να ε, κινηθεί με βάση την αγορά αυτή η προσπάθεια. Δεν μπορούμε να, ε, να επικεντρωθούμε μόνο σε μια ενδεχόμενη φούσκα που θα μπορούσε να δημιουργηθεί. Πρέπει να είναι κάτι βιώσιμο. Έχουμε βέβαια μια τέτοια αγορά στην Ευρώπη και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και οι πολιτικές σε εθνικό επίπεδο τη χάνουν συντονισμού και κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Αν έχουμε ένα προϊόν, ένα όχημα το οποίο ε, πωλείται υπό 27 διαφορετικά συστήματα και όρους, τότε αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και από πλευρά ε, επιτροπή η μεγάλη συμβολή είναι οι υποδομέ και τα πρότυπα. Εκεί πρέπει να γίνει η μεγαλύτερη προσπάθεια πρέπει ε, να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ κρατών μελών. Ιδίω, ας πούμε, είναι κάποιο εδώ στο Βέλγιο. Έχουμε, ε, συνορεύει Μεγαλία, Γαλλία, Ολλανδία και Γερμανία. Θέλει κάποιο να έχει ένα ηλεκτρικό όχημα, αλλά τι να κάνει. Υπάρχουν διαφορετικέ ε, προσεγγίσεις και συστήματα σε όλα αυτά τα αλλά δεν λειτουργεί. Μετά, ποιότητα καυσίμων που ορίζεται αρκετά καλά σε ό,τι αφορά τα ε, συνήθη αλλά για τα υπόλοιπα πρέπει να βελτιωθεί ο ορισμός. Υπάρχουν πολλές διατάξεις για, το, ε, για τους σταθμούς ε, ανεφοδιασμού και για το φυσικό αέριο και το καθεξής. Πρέπει να υπάρχει τυποποίηση και εκεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και για μας και για τους ε, καταναλωτές, τους πελάτες. όλη αυτή η προσπάθεια θα εξαρτηθεί από, την από τις υποδομές κατά τη γνώμη μας. Γι' αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε στις επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα. Και αυτό είναι ε, θέμα δράσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση, σίγουρα όμως και σε επίπεδο κρατών μελών. Ε, σίγουρα δεν είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος, όμως θα πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις και σε διάφορα εναλλακτικά καύσιμα. Ε, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, υγραέριο και το καθεξής. Τώρα, για την ηλεκτρική ενέργεια και, τον, και την επαναφόρτιση. Ξέρετε ότι όλοι συμφώνησαν, όλοι οι κατασκευαστέ συμφώνησαν πριν από ένα χρονικό διάστημα για τον τρόπο, που θα παράγουν οχήματα στο μέλλον. Συμφωνήσαμε ότι θα τυποποιήσουμε ε, το, την κατεύθυνση αυτή μέχρι το 2017 για τα νέα οχήματα, για τον τύπο 2 και τύπο 2 και έχουμε δεσμευτεί και προς τις ε, δημόσιες αρχές. Όμως πρέπει να τονίσουμε ότι χρειάζεται και μια μεταβατική περίοδος. Δεν θα γίνουν όλα μέσω του τρόπου 3. Πρέπει να δίνεται και δυνατότητα επαναφόρτησης και στο σπίτι και με διαφορετικούς τρόπους. Και σίγουρα πρέπει να υπάρχει συμβατότητα και με τα οχήματα που ήδη επαναφορτίζονται σήμερα. Κάμπος αυτό θα πρέπει να ε, διευθυντηθεί για το μέλλον. Όμως έχουμε ένα ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον. Τύπος 2 και τύπος 2 κόμπο λοιπόν. Λοιπόν, για την ε, καθαρή ενέργεια για τις μεταφορές, αυτό το πακέτο σίγουρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να βρούμε τρόπους να αποφευχθεί ο κατακαιρματισμός αγοράς. Πλέον έχουμε 27 διαφορετικές αγορές για τα τρένα εναλλακτικών καυσίμων και ούτω καθεξής, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Χρειαζόμαστε γρήγορα λύσεις που θα ωφελήσουν εξαιρετικά και τον κλάδο, γιατί υπάρχει εξοικονόμηση δαπανών, αλλά σίγουρα και πιο σημαντικό είναι ότι θα ωφελήσει και τους ε, πελάτες και θα τους βοηθήσει να επιλέξουν ε, οχήματα εναλλακτικών καυσίμων. Έχουμε ήδη λοιπόν συμφωνήσει για κάποια τμήματα Υπάρχει ήδη επιλογή, υπάρχει λοιπόν η λύση, τώρα πρέπει να λάβουν δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε. Κύριος Φιντάντζα. Μάισνερ, Τέιλορ, Λίχτενμπέργκερ και Κόλιτσεκ. Απλώς λέω ποιους έχω μέχρι στιγμής. Κυρία Φώστερ, γιατί όσο πιο πολύ μιλάμε, τόσο πιο λίγοι θα έχουν το λόγο, ο κύριος Γκρός επίσης, βεβαίως. Αυτή. Κύριε Έρτου και σας σας έχω βάλει. Ο κύριος Φιντάντσα. Οκτώ. Τρία λεπτά στον κύριο Φιντάντσα ως εισηγητή και δύο λεπτά στους άλλους. Πάμε. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι ακόμα πιο λακωνικός, διότι δεν ήθελα να κάνω παρέμβαση, απλώς κάποιες διευκρινήσεις ήθελα από κάποιους από τους ομιλητές, τους οποίους να ευχαριστήσω και παρεμπιπτόντως. Στον κύριο Κρίστη καταρχάς. Όσον αφορά το θέμα του εξηλεκτρισμού, εμείς στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων που κάναμε εδώ στην Επιτροπή μας, είχαμε πολλές παρεμβάσεις από πλευρά συναδέλφων για το θέμα της χρηματοδότησης διότι βεβαίως όλοι συμφωνούμε ότι πηγαίνουμε προς μια σωστή κατεύθυνση, προβλέπονται και μια σειρά από επενδύσεις ε, οι οποίες όμως ε, δεν είναι δυνατόν να το πιστούν από τον δημόσιο κορβανά. Πώς μπορεί λοιπόν να υπάρξει σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα ώστε να αποφύγουμε στο μέτρο του δυνατού τις επενδύσεις από πλευράς δημοσίου τομέα. Τώρα, όσον αφορά την πτυχή του φυσικού αερίου προς τον κύριο Μέτς, θα ήθελα μία διευκρίνηση για το κατά πόσον υπάρχει συμβατότητα μεταξύ υπεπιεσμένου φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Είδαμε κάποιες διαφάνειες, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσατε ίσως να μας εξηγήσετε λίγο καλύτερα τι γίνεται σε επίπεδο αποθήκευσης και διανομής. Μπορούν να συνδυαστούν αυτές οι δύο τεχνολογίες. Ε, και πάλι προς τον κύριο Μέτζ, ε, τι γίνεται με τους χιλιομετρικούς στόχους. Εσείς ε, θεωρείτε δηλαδή ότι οι χιλιομετρικοί στόχοι, η απόσταση μεταξύ των διαφόρων σταθμών ανεφοδιασμού είναι στόχοι τους οποίους μπορούμε να επιτύχουμε και ή μπορούμε να τους βελτιώσουμε και αν ναι προς ποια κατεύθυνση. Και μία ερώτηση και στον κύριο ε, Ρικό τη CV Plug Alliance. Μπορεί και να έκανα λάθος εγώ και να χάθηκα κάπου. Δεν κατάλαβα αν εσείς έχετε κάποια συγκεκριμένη θέση ως Plug Alliance για το θέμα ε, κόμπο 2 ή σαν σαντέμο. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο καλύτερα το σημείο αυτό. Ευχαριστώ κύριο Σέρτογκ και δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω δύο ή τρία συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα για τον κύριο Χρήστη. Είπατε ότι η πρίζα υπαριθμών 2 θα πρέπει να είναι το πρότυπο και είπατε επίση ότι οι άλλες μορφές ε, υποδοχών και πριζών δεν πρέπει να αποκλειστούν βέβαια, αλλά μήπως προτείνεται κάποιον ε, μετατροπέα ο οποίος θα μπορέσει να επιτρέψει τη χρήση και των δύο μορφών πρίζας. Δεύτερη ερώτηση προς την Κομισιόν και τον κύριο Σε ποιο βαθμό ε, αναρωτιέμαι για το εφικτό εδώ. Αναρωτιέμαι για το εφικτό σε ό,τι αφορά τη χωροταξία. Η κάθε χώρα έχει διαφορετικές δομές χωροταξίας, διαφορετική νομοθεσία. Πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό να πείτε ότι στις αστικές περιοχές, σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συγκοινωνίες, να έχουμε μεγαλύτερες δυνατότητες ε, για επαναφόρτιση, όλα αυτά τα βλέπω πολύ δύσκολα να τα εναρμονίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ένα ακόμα ερώτημα, τέλος, για τον κύριο Μέτς. Δεν κατάλαβα πολύ καλά. Μιλήσατε και για τη χρήση του μεθανίου μαζί με το πεπιεσμένο φυσικό αέριο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Μπορείτε να μας πείτε αν μπορεί να παράγεται αυτό το φυσικό αέριο, το υγροποιημένο, το πεπιεσμένο επί τη βάση μεθανίου ή όχι. Άλλο ένα ερώτημα είχα, τελευταίο, σε εσά κύριε Μέτς. Μιλήσατε για συνειδητοποίηση από την πλευρά του καταναλωτή. Με ποιο συγκεκριμένο τρόπο θα μπορέσετε να προωθήσετε αυτήν την ε, συνειδητοποίηση από την πλευρά του πολίτη και να την ενισχύσετε. Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ δεν θα τα χρησιμοποιήσω. Θέλω απλώ να ευχαριστήσω για τις παρουσιάσεις. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. <clears throat> Βλέπω ότι υπάρχει γενική συνένεση για την πρόταση αυτή. Το θέμα των ε, μετατροπέων ή των ε, πριζών νομίζω ότι έχει ε, διευκρινιστεί. Δύο ερωτήματα, πρώτα για τον κύριο Τσίολεκ για το πεπιασμένο και το εγροποιημένο φυσικό αέριο. Μιλήσατε για τα κίνητρα τα οποία πρέπει να, έχουν, υπάρχουν για τις περιφέρειες. Πιστεύετε τώρα ότι αυτή η πρόταση λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά κίνητρα που υπάρχουν από τις περιφέρειες και επίσης δημιουργία υποδομής για μεθάνιο. Το άλλο ερώτημα αναφέρεται στον κύριο Ντολέση, ελπίζω ότι δεν κακοποιώ το όνομά σας, σε σχέση με τις επενδύσεις. Ίσως είναι κρίσιμο το ερώτημα αυτό. Εσείς με τη δική σας εμπειρία και με τις επαφές που έχετε θεωρείτε ότι υπάρχει επαρχή συνειδητοποίηση για τα θέματα αυτά. Υπάρχει κάτι λοιπόν το οποίο μπορείτε να διευκολύνετε με τη δική σας δράση. Ο κύριος Τέιλα. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους για τις παρουσιάσεις σας. Δύο σχόλια μονάχα. Για μένα τα ηλεκτρικά οχήματα δεν είναι μια σοβαρή επιλογή για ένα γιοταχή, γιατί έχουν περιορισμένη εμβέλεια μέσα στην οποία μπορούν να κινηθούν. Μιλάω για καθαρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όχι υβριδικά. Δεν μπορούν να πάνε πολύ μακριά. Και αυτό δεν βολεύει πολλούς χρήστες. Για να παίξουν το ρόλο του κυρίου του οχήματος. Ο αντίκτυπος στο, σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος και τα πλεονεκτήματα της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων υπονομεύονται εκτός αν η παραγωγή ηλεκτρισμού έχει γίνει από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό όμως δεν το αναφέρετε στην παρουσίασή σας. Ή αν το παρουσιάσατε εγώ δεν το πιασα. Το θέμα εδώ είναι ότι οι επενδύσεις και η προτυποποίηση χρειάζονται και για τα ηλεκτρικά οχήματα και για τα οχήματα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Και αναρωτιέμαι αν είναι ίσως κάπως πρόορη αυτή η κίνηση για την προτυποποίηση, γιατί το πεπιεσμένο φυσικό αέριο και το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι ένας πόρος ο οποίος είναι πεπερασμένος. Ενώ η δημιουργία υποδομών οδηγεί σε τεράστιο κόστος. Θα σας ενθάρρυνα λοιπόν να συνεργαστείτε περισσότερο με την αυτοκινητοβιομηχανία για να παραγάγουν οχήματα τα οποία πράγματι θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν οι καταναλωτές. Κύριε Λίχτεμπερ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να θέσω κάποια μικρά ερωτήματα. Παρακολούθησα τη συζήτηση για τη δημιουργία προτίμων την έχω παρακολουθήσει εντατικά. Βλέπω τώρα ότι υπάρχει και μία σύγκρουση μεταξύ των δύο προτύπων. Έχουμε ένα βασικό πρόβλημα. Εάν κάνω πρόορη προτυποποίηση, αποκλείω την καινοτομία, η οποία μπορούσε να φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Εάν καθυστερήσω την προτυποποίηση, τότε έχω ένα μεγάλο αγώνα μεταξύ των υποδειγμάτων που υπάρχουν που δεν μπορώ να τον διαλευκάνω. Ποια είναι η θέση σας για τα θέματα αυτά. Το θέμα της προέλευσης συνεργητικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στα ηλεκτρικά οχήματα αναφέρθηκε ήδη από τον κύριο Τέλο. Εγώ θέλω να προχωρήσω λίγο περισσότερο όμως. Όταν δω <clears throat> τα θέματα εφαρμογής, παραδείγματος χάρη, την ηλεκτρική κινητικότητα. Δεν είναι μόνο το θέμα των μεταφορών μεγάλων ε, αποστάσεων που πλήττεται από την περιορισμένη εμβέλεια, και δεν πρέπει να δημιουργήσουμε ψευδεστήσει στους πολίτες. Αλλά πράγματι όπως ελέγχθη, τι θα κάνω στις πόλεις. Υπάρχει το θέμα της χωροταξία. Πρέπει να δημιουργήσω χώρους επαναφόρτηση των ε, οχημάτων. Σε περιοχές της Υπέθρου αυτό δεν είναι δύσκολο. Αλλά πού θα βρούμε χώρο να φτιάξουμε τα γκαράζ για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στι πόλει Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και τέλος, με ποιο τρόπο θα μπορέσει να γίνει η εφαρμογή στου τομείς αυτού. Βλέπω να είναι πολύ δύσκολα όλα αυτά. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο λοιπόν η προσβασιμότητα στις αγροτικές περιοχές αλλά στις πόλεις. Και υπάρχει και το θέμα της περιορισμένης ακτίνας δράσης για τα οχήματα τα ηλεκτρικά. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές από όλα αυτά τα οποία παρουσιάζονται στις διαφημίσεις για τα ηλεκτρικά οχήματα. Λαμβάνει κανεί υπόψη την απόσταση που μπορεί να διαθέξει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο άμα δεν χρησιμοποιείται καθόλου ηλεκτρική ενέργεια στο αυτοκίνητο, παραδείγματο χάρη ραδιόφωνα ή συστήματα πλοή κτλ. Αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Κόλλησε πια δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας πω ότι θεωρώ ότι οι συνάδελφοι αναμειγνύουν δύο πράγματα. Εγώ σπούδασα χημεία και πιο συγκεκριμένα η διπλωματική μου εργασία αφορούσε θέματα ε, ε, που έχουν σχέση με τη δημιουργία θερμότητας και κάθε φορά που δημιουργείται θερμότητα ε, υπάρχουν και κατάλοιπα διοξιδίου του άνθρακα. Θεωρώ λοιπόν ότι τα αέρια στα οποία αναφερθήκατε εσείς ή μπορούν να προκύψουν από το υδρογόνο που θα ήταν και το ιδεώδες φυσικά. Ε, υπάρχουν ίσως και οι δυνατότητες ε, χρήσης άλλων ε, ε παραγωγής τους από άλλες δυνατότητες, αλλά θα ήταν πιο περίπλοκα. Θα μπορούσε ίσως να υπάρχει και κάποιος συνδυασμός χρήσης καυσίμων στα αυτοκίνητα οχήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις... δεν εξετάζεται καθόλου με ένα, αλλά υπάρχουν χώρες στις οποίες εξετάζονται κάποιες εναλλακτικέ λύσεις. Το θέμα είναι τι είδου ε, φόρτιση θα έχουμε, 220 βολτ, 360, ε, πώς θα γίνεται η ηλεκτρική φόρτιση, τι είδους βίσμα θα χρησιμοποιείτε και ε, η άλλη με ερώτηση είναι η εξή. Έστω ότι έχω μια μπαταρία την οποία μπορώ κάλλιστα να την αποσυνδέσω ε, και να αφαιρέσω τελείω την μπαντερία, να την επαναφορτήσω ξεχωριστά και να την επανατοποθετήσω στο όχημα. Αυτό ε, ίσως ε, θα διευκολύνει κάποιες διαδικασίες διότι δεν θα υπήρχε άλλη επιβάρυνση και θα μπορεί να γίνεται ξεχωριστή επαναφόρτιση ε, με την ίδια μπαταρία. Επίσης, αν θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε και συγκεκριμένους σταθμούς επαναφάρτησης ή συγκεκριμένα ε, εξαρτήματα τα οποία θα ε, παρασκευάζονται ευθύς εξ αρχή ώστε να χρησιμοποιούν καθαρή ενέργεια το οποίο ναι θα κοστίσει λίγο περισσότερο αλλά θα είναι πιο αποδοτικό στη συνέχεια. Κυρία Φώστερ, ευχαριστώ πολύ. Θα έπρεπε να ήμουν πιο επιμελής και εγώ στα μαθήματα χημίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κόλιτσεκ που μας δώσατε λίγες ε, ε, πληροφορίες, μια χτίδα φωτός για το πώς ε, λειτουργεί αυτό το σύστημα. Νομίζω ότι όλοι καλωσορίζουν το γεγονός ότι ε, μπορούμε να χρησιμοποιούμε εναλλακτικέ πηγές καυσίμων και ούτω καθεξής. Να υπενθυμίσω βέβαια στους δύο ομιλητές ε, ως ε, κλάδος ή ως βιομηχανία ή ως μη κυβερνητική οργάνωση ή οποιοδήποτε άλλος δεν καταθέτετε εσείς τροπολογίες. Αν είναι κάποιο να υποβάλει τροπολογίες, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αυτά τα οποία αποφασίζουν τι θα κάνουμε την νομοθεσία. Θα ήθελα να στο υπενθυμίσω με κάθε ε, ευγένεια. Ήταν ενδιαφέρουσες βέβαια η παρουσιά σας, αλλά δεν νομοθετείτε εσείς. Νομίζω ότι το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει χρονοδιαγράμματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν ναι μεν υπάρχει ένα στόχος, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν μπορεί να γίνονται αυθαίρετα πράγματα για κάτι τόσο περίπλοκο όπως είναι το συγκεκριμένο ζήτημα. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να θέσουν στόχους, γιατί είναι πολύ δύσκολο να θέσουν στόχους ούτως ή άλλως. Και ε, εδώ συμφωνώ με την αυτοκινητοβιομηχανία. Υπάρχουν αυτοκινητοβιομηχανίες και στη δική μου την περιοχή και σε όλη την Ευρώπη, ότι όλα αυτά ε, εξαρτώνται από την αγορά. Μόνο αν καταναλωτής επιθυμεί κάτι ή όχι και οι ε, αυτοκινητοβιομηχανίες μπορούν να τους ε, κατασκευάσουν κάτι που επιθυμούν είναι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει. Υπάρχει και ένα θέμα επικουρικότητα εδώ. Κατά την άποψή μου Πρέπει να δούμε και τι θα αποφασίσουν να κάνουν τα κράτη-μέλη, διότι βλέπουμε και πώς είναι η γεωγραφία μιας χώρας. Εξετάζουμε και άλλους παράγοντες για να δούμε αν ένα κράτος μέλος θα αποφασίσει να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Και αυτό που δεν ανέφερε κανείς είναι το κόστος των υποδομών δεν είναι ε, χωρίς κόστος, δεν έρχεται δωρεάν αυτή η υποδομή. Ίσα ίσα είναι τεράστιο το κόστος για να ε, κατασκευάσουμε υποδομές που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουμε τα θέματα αυτά. Ίσως σε μια επόμενη συνεδρία θα το συζητήσουμε, αλλά το πάνελ το απέκρυψε ε, εντελώ και είναι και ένα από τα πιο σημαντικά θέματα και θα είναι και ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για τα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν. Μας ενδιαφέρει συνεργασία λοιπόν μεταξύ κυβερνήσεων και του κλάδου φυσικά ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο να είναι λίγο πιο λογικό από αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Και τέλος, ο κύριος Γκρός για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τις, τους εμπειρογνώμονες για τις τόσο ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Ξέρουμε ότι τα επόμενα χρόνια ο 80% του πληθυσμού θα ζουν στις πολίτες και εδώ τίθεται το θέμα της χρήσης των συγκοινωνιών στις πόλεις και τις αυτονομίες που έχουν. Στις Βρυξέλλες λέει μια μελέτη ότι θα περάσουν σε ηλεκτρική κινητικότητα τα 50% των κατοίκων, αλλά δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές για αυτό το πράγμα. Πώς λοιπόν θα τοποθετηθείτε για αυτό το θέμα, πώς θα αντιμετωπιστούν οι ανάγκες όταν είναι μια πολύ γρήγορη ανάπτυξη ηλεκτρικής κοινωνικότητας. Επίσης, η προτυποποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Όταν εγώ πηγαίνω σε μικρές αποστάσεις, βέβαια δεν είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με αυτονομία, αλλά χρειάζεται πράγματι να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα ή μήπως και οι ίδιες οι βιομηχανίες ηλεκτρικών οχημάτων ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν αυτή την διαλειτουργικότητα για να μπορέσουν να έχουν μεγαλύτερη ε, ελκυστικότητα για τους καταναλωτές. Είχαμε πολλά προβλήματα που έχουμε δει σε σχέση με τις τεχνολογίες γιατί δεν υπάρχουν συμβατές τεχνολογίες και έπρεπε η ίδια η βιομηχανία να τα ρυθμίσει. Τέλος έχω το θέμα της ασφάλειας. Παραδείγματος χάρη όταν έχουμε τώρα μεγάλα γκαράζ τα οποία έχουν αυτοκίνητα με φυσικό αέριο. Χρειάζεται κάποιο είδος ειδικών υποδομών και επίσης οι υποδομές επαναφόρτισης στον χώρο των πόλεων. Αυτό το θέμα δεν έχει επιλυθεί ακόμα. Αυτά είναι θέματα λοιπόν τα οποία τα ενδιαφέρουν τους καταναλωτές. Πρώτον η τιμή, δεύτερον η προτυποποίηση, τέταρτον η ασφάλεια και μετά η αυτονομία. Αυτά είναι τα θέματα που δείχνουν δημοσκοπήσεις ότι θέλουν οι καταναλωτές να είναι σε θετική κατάσταση για τα ηλεκτρικά οχήματα. Ευχαριστώ. Κοιμάστε. Ναι. Πρέπει να πάω σε μια άλλη επιτροπή και δεν είναι ευγενικό να θέτω ένα ερώτημα και να φύγω. Αυτό, αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, θα ήθελα να το επισημάνω στους εισηγητές μας. Και κάποιος που δεν έχει πολύ καλές σημειώσεις για τα θέματα χημίας και φυσικής και κάπου δημιούργησα μια μικρή έκρηξη όταν ήμουνα 11 χρονών. Ξέρω ότι έχετε πίεση χρόνο αλλά μπορείτε πάντα να δώσετε και έγγραφες απαντήσεις στα μέλη. Δύο λεπτά, κύριος Χρήστης πρώτος. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισμένα ερωτήματα για τη χρηματοδότηση υπάρχουν πολλά επιχειρηματικά πρότυπα που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Υπάρχουν κάποιες δυνατότητες και ευκαιρίες ε, όταν έχουμε επενδύσεις για τις υποδομές, μετά κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο. Υποδομές λοιπόν μαζί με ένα εμπορικό ε, κατάστημα που ε, προσελκύει πελάτες, καταναλωτές και έτσι έχουμε ένα ευρύτερο πακέτο ή επιχειρηματικά μοντέλα όπως με το σύστημα κινητής τηλεφωνίας, με δυνατότητες ε, περιαγωγής. Το βασικό είναι να μην υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις, πολλοί... οι τροπολογίες ανέφερε ο μιλήτης, μάλλον οι προτάσεις μας για τροπολογίες που θα καταθέσουν οι ευρωβουλευτές προβλέπουν ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν πολλοί περιορισμοί ε, για τον τρόπο επένδυσης. Να μην εμποδίσουμε λοιπόν κάποια επιχειρηματικά ε, μοντέλα, αλλά μπορούμε να το τεκμηρέσουμε περαιτέρω αυτό που σας λέω. Για τον κύριο Τέιλορ, και αυτό συνδέεται και με τα όσα είπε ο κ. Γκρό στο τέλος είναι ακριβώς αυτό που αφορά τις ε, χώρες όπως την Ευρώπη με μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα κτλ. Ε, υπάρχει μεγάλη μετακίνηση σε μικρές αποστάσεις, επομένως μεγάλο τμήμα του πληθυσμού θα μπορούσε πολύ εύκολα να ε, περάσει στην ε, ηλεκτροκίνηση, ιδίω αν αυτό συνδέεται και με τις δημόσιες μεταφορές. Δεν είναι για όλους, ούτε για όλες τις μορφές μεταφορών. Δεν είναι καλό πούμε, για τις καλοκαιρινές διακοπές, προφανώς. Αλλά σίγουρα σε ένα βαθμό μπορεί να λειτουργήσει. Και πράγματι στις αστικές περιοχές ε, υπάρχει και το ζήτημα της συμφόρησης. Γι' αυτό και έχουμε αυτή την πολυτροπική πλατφόρμα. Δεν θα αντικαταστήσουμε όλα τα συμβατικά οχήματα με ηλεκτρικά. Ευχαριστούμε. Βεβαίως και μπορείτε πάντα να απαντήσετε και γραπτώς ε, στα μέλη του Κοινοβουλίου. Κύριος Μάτζ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Φώστερ, βεβαίω δεν έχω ε, καμία πρόταση για τροπολογίε. Εμεί απλώ σα λέμε τι δικέ μα απόψει επί του θέματο. Προφανώς δεν υπάρχει σημαντικό ζήτημα για το φυσικό αέριο στην πρόταση, γιατί έχει οριμάσει και η τεχνολογία. Να απαντήσω στα ερωτήματά σας πριν να απαντήσω στον κύριο Φιντάντσα. Τι είναι το πεπιεσμένο και το υγροποιημένο είναι μεθάνιο. Ναι, πράγματι το ε, πεπιεσμένο και το υγροποιημένο πάντα ε, μιλάμε για το ίδιο καύσιμο. Δεν πρέπει να το ε, συγχέουμε με το LPG, το υγραέριο. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Άλλο το CNG και το LNG που είναι μεθάνιο, φυσικό αέριο πλούσιο σε μεθάνιο και μπορεί να είναι είτε ορυκτό είτε ανανεώσιμο. Η τεχνολογία είναι απόλυτα συμβατή, κύριε Φιντάντσα, και μπορείτε να τη συνδυάσετε. Μπορούμε να συνδυάσουμε και τι δύο τεχνολογίε η βασική διαφορά είναι η αποθήκευση. Το φυσικό αέριο γίνεται υγροποιημένο όταν ε, ψυχραίνεται στους 160 βαθμούς και τότε καταλαμβάνει λιγότερο χώρο. Σε ένα όχημα λοιπόν όπου χρησιμοποιούμε πεπιεσμένο φυσικό αέριο, προφανώς δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το, ε, να χρησιμοποιήσουμε το LNG, γιατί αν πάει κάποιες δικοπές και αφήσει το ε, όχημά του σπίτι, τότε αυτό εξαερώνεται μετά από μια-δύο εβδομάδες. Επομένω με το LNG πρέπει κάποιο να το χρησιμοποιεί αμέσω, ε, συνέχεια. Οι υποδομέ ε, και πάλι είναι, η διαφορά είναι σύνδεση με, τη, τον αγωγό είτε η χρήση μια δεξαμενή. Ο χιλιομετρικό στόχο, κύριε Φιντάντσα, βεβαίω και μπορεί να βελτιωθεί. Πολλοί λένε τα 150 να γίνουν 50, τα 400 να γίνουν 200 αλλά τα 400 και τα 200 βασίζονται σε συγκεκριμένες προοπτικές και συγκεκριμένους στόχους μπορεί να πετύχει το κάθε τύπο οχήματος. Πώς μπορούμε να κινήσουμε το ενδιαφέρον των καταναλωτών. Αυτό αφορά και την διάρκεια ε, της ε, μετακίνησης ε, και το θέμα της τιμής Ναι, συγγνώμη που μακρηγορώ. Βεβαίω και είναι πεπερασμένο φυσικό πόρο. Κάποια στιγμή θα τελειώσει, αλλά είναι σε αυθονία. Και γι' αυτό πρέπει να ε, αξιοποιήσουμε αυτό το φυσικό πόρο. Αυτά ήθελα να πω. Ναι, συγγνώμη, πρέπει να σας διακόψω, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Ζιόλεκ, παρακαλώ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Δύο σχόλια έχω. Για τα κίνητρα μπορούν να δοθούν σε τοπικές αρχές και περιφέρειες για την επίτευξη των στόχων της οδηγία. Προ το παρόν ε, είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι σε ό,τι αφορά ε, τις εξελίξεις. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων. Από τα αποτελέσματα που βλέπουμε μέχρι σήμερα βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Και αυτό ακριβώ θα θέλαμε να τονίσουμε και να ενδυναμώσουμε αυτό το στοιχείο στο μέλλον. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις υποδομές και πώς οι υποδομές ε, ηλεκτροκίνηση μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ε, πρέπει να συνδυάσουμε όλες τις μορφές ηλεκτρικών ε, οχημάτων. Δεν μπορώ να σας δώσω δυστυχώ μία και μοναδική απάντηση, γιατί υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ε, και διαφορετικά συστήματα. Άλλη κατεύθυνση ακολουθεί το Όσλο, άλλη το Παρίσι. Αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Βασική κινητήρη μοχλή σε ε, περιφερειακό, περιφερειακό επίπεδο είναι η ενσωμάτωση των νέων φορέων παροχής που θα πρέπει να ενταχθούν στη διαχείριση του δικτύου. είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή και για, τις, ε, για τους τοπικούς φορείς. Ε, κύριε Ρίκο. Υπήρχε μια ερώτηση από τον κύριο Φιντάντσα για το τι άποψη έχουμε για το κόμπο 2 και το σαντεκό. Αυτό έχει σχέση με την ε, σύνδεση στο αυτοκίνητο. Επομένω, μάλλον ο συνάδελφο θα μπορούσε να απαντήσει. Η θέση μα είναι όμω ότι δεν θα πρέπει να τιμωρούμε του καταναλωτέ που έχουν ε, ε, ήδη αυτοκίνητα με το σύστημα σάντεμο και επίση η ταχεία επαναφόρτωση ε, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αποδοτική. Εμεί θεωρούμε ότι τα περισσότερα οχήματα θα πρέπει να, είναι, ε, να έχουν τη δυνατότητα μια ημιταχεία επαναφόρτηση στα 22 χιλιόμετρα. Επίση, η ευφυή επαναφόρτηση είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι θα μα επιτρέψει να έχουμε μεγάλη δυνατότητα χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργεια. Θα μπορούσα να σα δείξω ένα παράδειγμα. Το μεγαλύτερο τμήμα του αυτοκινήτου θα περιλαμβάνει επιπλέον ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα παράγονται από ανεμόμυλους όταν δεν θα μπορεί να καταναλωθεί ενέργεια. Δηλαδή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να αποτελέσει και λύση στο πρόβλημα και όχι ε, πρόβλημα για τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υπήρχε και μια ερώτηση για το κόστος των υποδομών. Εδώ θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε ε, όσο το δυνατόν περισσότερες δυνατότητες επαναφόρτησης σε κτίρια και σε κατοικίες, ε, όπου το κόστος θα είναι πολύ λιγότερο από την εγκατάσταση υποδομών ε, στα πεζοδρόμια, όπου θα χρειάζεται και δημόσια επένδυση. Και υπήρχε και μια ερώτηση για τις πόλεις στις πόλεις ε, θα είναι πολύ σημαντικό το μοντέλο του car sharing, το να μοιράζεται κάποιος ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ε, η ηλεκτρική χρήση αυτοκινήτων σημαίνει και νέες αντιλήψεις ε, για χρήση και επαναφόρτιση. Δεν σταματώ για να επαναφορτήσω, επαναφορτήσω γιατί σταματώ και πρέπει να χρησιμοποιούμε λοιπόν τις υποδομές σε σταθμούς στους οποίους θα πρέπει να σταματήσει κάποιο το αυτοκίνητό του για 50 λεπτά ή 8 ώρες και να προσταρμόσουμε την απόδοση βάσει αυτό και φυσικά είναι απαραίτητο να υπάρχει ε, κατά νου συνέχεια η ασφάλεια. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά μας πριν εγκριθεί οποιαδήποτε ε, οδηγία. Και τέλος, ο κύριος ε, Ντολιέση, θα ξεκινήσω από τα τελευταία σχόλια του κυρίου Γκρός. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μία λύση για την Ευρώπη. Είναι γελίο να είμαστε παγκόσμιε επιχειρήσει ε, οι οποίε μπορούν να πολλούν αυτοκίνητα στι Ηνωμένε Πολιτείε, στην Κίνα και να μην μπορούμε να πολλούμε τα ίδια αυτοκίνητα στη Γαλλία και στη Γερμανία. Λυπάμαι πολύ που το λέω έτσι. Μα ικανοποιεί ιδιαίτερα λοιπόν το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια λύση για την Ευρώπη και να φτάσω και στην ερώτηση τη χρηματοδότηση. Εμεί δεν ζητάμε να γίνουν επενδύσει δισεκατομμυρίων, ζητάμε μια επένδυση προ την ίδια κατεύθυνση. Να υπάρχει εξορθολογισμένη και εναρμονισμένη επένδυση σε μια συγκεκριμένη λύση. Ειλικρινώς να σας πω ότι στην πρώτη διαφάνεια είδατε ότι οι πελάτες μας επενδύουν ετησίως 26 δισεκατομμύρια ευρώ ε, ε, για έρευνα και καινοτομία. 26 δισεκατομμύρια για λύσεις οι οποίες ε, μπορεί και να μην είναι αποδοτικές και μπορεί να είναι και επιχειρηματικός κίνδυνος. Ε, δεν μπορούν να μας λένε τα κρατημέλη λοιπόν ότι θα πάμε προς μια κατεύθυνση και μετά συγγνώμη δεν θα σας δώσουμε ούτε δεκάρα τσακιστή. Λυπάμαι πολύ αλλά δεν είναι σωστή αυτή η προσέγγιση. Σας λέμε λοιπόν ότι αναλαμβάνουμε εμεί τον κίνδυνο, χρησιμοποιούμε διάφορες δυνατότητες και παράγουμε και διαθέτουμε προϊόντα στην αγορά. Επαφίεται λοιπόν τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη να κάνουν και αυτοί το μερίδιό τους στην επένδυση. Γνωρίζετε επίσης ότι τα μισά κράτη-μέλη τουλάχιστον έχουν εθνικά σχέδια. Ε, υπάρχει ε, σχέδιο Γαλλία, Δανία, Γερμανίας για την ηλεκτρική κινητικότητα, αλλά κατασπαταλούνται χρήματα σε διαφορετικές λύσεις. Εμείς δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε τα κράτη-μέλη, θέλουμε να υπάρχει ένας εξορθολογισμός, να πάμε προς μία κατεύθυνση, να συμφωνήσουμε, να πούμε θα πάμε προς αυτή τη μεριά και να επενδύσουμε όλοι προς αυτή. Και νομίζω ότι και αυτοί που παρέχουν τι υποδομές ευχαρίστως ε, θα μοιραστούν τους πελάτες τους μαζί μας. Αν έχουμε λοιπόν μια κοινή προσέγγιση και να μοιραστούμε ο καθένα το μερίδιό του του κόστου και πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια λύση για την Ευρώπη. Ευχαριστώ, να ευχαριστήσω όλου του εμπειρογνώμονε λοιπόν από το πρώτο πάνελ και να περάσουμε τώρα στο δεύτερο πάνελ. Ε, να αλλάξουμε λοιπόν θέσει για να περάσουμε στη δεύτερη βάρδια. Το δεύτερο πάνελ περιλαμβάνει τον κύριο William Λάρος από τις υδατόβιες τεχνολογίες, τον κύριο Μπιγιέτ από την ε, Παγκόσμια Ένωση Οδικών Μεταφορών, τον κύριο Ουμπέρτο από την Παγκόσμια Οργάνωση Δημοσίων Μεταφορών, την κυρία Σίλβεν Χάον από την πόλη στο δίκτυο των πόλεων και των περιφερών και τον κύριο Μαρίνο Μάρτενς από την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αν μπορείτε λοιπόν να έρθετε εδώ Καθίστε όπου θέλετε. Απλώς βρείτε μια θέση να κάτσετε. Okay, colleagues, are Πάμε συνάδελφοι λοιπόν, ξεκινάμε και πάλι. Οι ήδη κανόνε που εφαρμόζονται στο δεύτερο ημίχρονο όπως και στο πρώτο ημίχρονο θα είμαι αμήλικτος με τη χρήση του χρόνου. Έξι λεπτά λοιπόν ο κύριος Βίλεμ Λάρτς για τις υδατόβιες τεχνολογίες. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σας κύριε και κύριοι, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, για το γεγονός που μας δίνετε την ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί σας ορισμένες ιδέες από τον κόσμο των θαλασσίων τεχνολογιών. Η Waterborne είναι μια πλατφόρμα τεχνολογιών που περιλαμβάνει όλους τους ε, ε, κύριους εμπλεκόμενους στον θαλάσσιο χώρο, τους ναυτικούς, τους μηχανολόγους θάλασσας, τους εφοπλιστές, η χρήση των καθαρών καυσίμων είναι ένας πάρα πολύ νευραλικός τομέας έρευνας για μας μέσα στα πλαίσια της πλατφόρμας μας. Πάντα θέλουμε να έχουμε χαμηλότερη κατανάλωση, καλύτερα καύσιμα ή ακόμα και χρήση και μη χρήση καυσίμων. Και φυσικά μας ενδιαφέρει και όλη αυτή η τεχνολογία που θα βελτιώσει την ποιότητα των καυσίμων με φυσικό αέριο. Αυτή η τεχνολογία ανατρέχει στη δεκαετία του 60 όταν η μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων υγροποιημένου φυσικού αερίου έγινε ρουτίνα και πολλά πλοία χτιστήκανε με την ε, λογική του να χρησιμοποιούν ένα τμήμα του φορτίου τους για να μεταφέρουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Δημιουργηθήκαν λοιπόν τουρμπίνες που χρησιμοποιούσαν φυσικό αέριο και τον τελευταίο καιρό είδαμε να χρησιμοποιείται το υγροποιημένο φυσικό αέριο ή άλλα καθαρά καύσιμα σαν εναλλακτική λύση για τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα. Υπάρχει εδώ όμως ένα μεγάλο ερωτηματικό για τα καύσιμα. Πού θα τα αποθηκεύσουμε. Όπως ξέρετε το υγροποιημένο φυσικό αέριο πρέπει να αποδικαίωται σε θερμοκρασία με 160 βαθμών και πρέπει κανείς να έχει αρκετό φυσικό υγροποιημένο αέριο για να μεταφερθεί από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι περιορίζουμε τον χρήσιμο χώρο στα οχήματα. Γι' αυτό το λόγο η χρήση των καθαρών αερίων και στη συγκεκριμένη περίπτωση του υγροποιημένου φυσικού αερίου ως εναλλακτική λύση εστιάζεται μόνο στις ε, σύντομες θαλάσσιες μεταφορές και στην εσωτερική, ε, στις εσωτερικές διαδρομές μέσα σε εσωτερικούς υδάτινους δρόμους. Και εκεί υπάρχει η δυνατότητα βέβαια να ανα, ανεφοδιάσετε το σκάφος πιο συχνά. Όταν μιλάμε για σκάφη τα οποία κινούνται με φυσικό αέριο, σκέφτεται κανείς τα φέρι τα οποία κάνουν σύστημες, σύντομες διαδρομές, τα ρημουλκά, τα πλοία που κινούνται σε εσωτερικούς υδάτινους δρόμους, ιδίως μεταξύ πυκνοκατοικημένων περιοχών. τα κοινωνικά ωφέλη και το κόστος άμα περάσουμε σε μια τέτοια χρήση φυσικού αερίου, καταρχήν μειώνουμε τις εκπομπές και συμμορφωνόμαστε με τους κανονισμούς για το περιβάλλον. Κατά 90% η μείωση οξύδια του θείου, ε, συμμορφωνόμαστε με την ε, οδηγία για τις ε, εκπομπές οξυδίων του αζότου, μείωση 20-25% για το διοξείδιο του άνθρακο, άνθρακος και τα εναλλακτικά καύσιμο όπως είναι το υγροποιημένο φυσικό αέριο καλύπτουν τις προδιαγραφές για το δίζελ είναι πιο αποτελεσματικά σχέση με το δίζελ και καλύπτουν τις προδιαγραφές ε, και είναι πιο αποδοτικά σε σχέση με το, με το βαρύ αργό πετρέλαιο. Και βλέπετε ότι βελτιώνεται η κατάσταση και εδώ. Αλλά έχουμε ακόμα το πρόβλημα του όγκου που χρησιμοποιείται για το, για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, οπότε σε εμπορικό επίπεδο δεν έχουμε ακόμα ένα πλέον έκτημα. Και υπάρχει, όπως είπα, η εστίαση σε σύντομες μεταφορές. <clears throat> που είναι όμως σημαντικές και όπως αναφέρει πρόταση Κομισιόν. Προκλήσεις τώρα και δυσκολίες. Μία από τις μεγάλες λοιπόν προκλήσεις είναι ο ανεφοδιασ... ο... οι υποδομές ανεφοδιασμού. Η Κομψιό θα πρέπει να επιλέξει τους λιμένες όπου πρέπει να υπάρχει μια τέτοια υποδομή για φυσικό αέριο. Το υποστηρίζουμε αυτό. Ε, με την υπενθύμηση ότι η Κομισιό πρέπει να αφήσει και την ε, αγορά να λειτουργήσει. Επίσης, είναι απαραίτητο να κρατήσουμε ζωντανή την καινοτομία για την τεχνολογία. Δεύτερον, έχουμε πρόβλημα έλλειψης συγκεκριμένων κανόνων και εναρμονισμένων προτύπων για την, τον ανεφοδιασμό και την αποθήκευση του φυσικού αερίου σε πλοία. Ο Διεθνής Νομισμα... Ε, Ναυτιλιακός Οργανισμός λειτουργεί με ένα, αλλά λειτουργεί με αργούς ρυθμούς. Και εδώ υπάρχει μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλύψει τις σύντομες μεταφορές και τις ε, μεταφορές σε εσωτερικούς υδάτινους δρόμους που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προωθήσει τα καθαρά καύσιμα και τις υποδομές ανεφοδιασμού. Κλείνοντας, εμείς υποστηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία και υπάρχει και μια πραγματική ευκαιρία να επιδείξουμε την ικανότητα των σημερινών τεχνολογιών να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στις θαλάσσιες μεταφορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λάρος. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Μαγμπιλιέτ από την ε, Διεθνή Ένωση Οδικών Μεταφορών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν υπάρχει λόγος βεβαίως να σας παρουσιάσω και πάλι την ένωση την οποία εκπροσωπώ. Θα περάσω λοιπόν κατευθείαν στο ουσιαστικό κομμάτι της παρουσίασής μου, το πακέτο για την καθαρή ενέργεια της μεταφορές. Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες της Επιτροπής ε, μέχρι τώρα. Οι εμπορικοί φορείς χρειάζονται ε, τα βιώσιμα εναλλακτικά καύσιμα για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας ίχνος στις οδικές μεταφορές. Αυτή η δέσμη, αυτό το πακέτο δείχνει ξεκάθαρες ε, εξελίξεις ε, και στις εμπορικές μεταφορές. Βελτιώνει ή θα μπορούσε να βελτιώσει τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών ε, καυσίμων σε διασυνοριακό επίπεδο. Μπορεί να παράσχει διαφανείς και αξιόπιστες πληροφορίες για την ε, αξιοποίηση αυτών των καυσίμων και θα μπορούσε να συμβάλλει στην επίλυση και αντιμετώπιση υφιστάμενων προκλήσεων. Ωστόσο, αυτό το πακέτο δεν μπορούμε να το εξετάζουμε μεμονωμένα. Είναι ένα κομμάτι ενός μεγαλύτερου πάζλ. Χρειαζόμαστε μια ολιστική προσέγγιση προς ε, το πρασίνισμα των μεταφορών. Δεν μπορούμε λοιπόν να εξετάζουμε μόνο τις υποδομές και τα καύσιμα, πρέπει να εξετάζουμε και τα οχήματα. Αυτό έχει ήδη αναφερθεί. Και οι φορείς μεταφορών θα πρέπει να ενθαρρύνονται, να παροτρύνονται να επενδύουν σε αυτά τα οχήματα. Και μετά είναι σημαντικός ε, με αξιόπιστο και διαφανές ε, τρόπο και διαφανή τρόπο να ε, βλέπουν τα ωφέλη αυτών των οχημάτων. Και τέλος, κυρίες και κύριοι, αυτός ο κύκλος που βλέπετε στο κέντρο, η χρηματοδότηση, ποιος θα πληρώσει και με ποιον τρόπο. Κάποιες από τις προκλήσεις τώρα. Δυστυχώς, μέχρι τώρα, αυτά τα οχήματα είναι ακριβότερα και στην πώληση και στην χρήση τους, την αξιοποίησή τους, σε σχέση με τα συμβατικά οχήματα υπάρχει και μια σύγκριση βάρους έναντι όγκου του ε, καυσίμου και του αντικτύπου στον, στη δεξαμενή. Και βλέπουμε ότι στην ε, υφιστάμενη πρόταση η Επιτροπή έχει λάβει υπόψη το ζήτημα των ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά όχι για τα υπόλοιπα ε, εναλλακτικά καύσιμα. Αυτό ίσως θα πρέπει να το εξετάσουμε. Άλλο θέμα είναι η αυτονομία ένα φορτηγό 40 τόνων με δίζελ κάνει 2.100 ε, χιλιόμετρα. Με υγροποιημένο κάνει μόνο 1.200. Μόνο με την ε, διπλή προώθηση ε, μπορούμε να αγγίξουμε ή να πλησιάσουμε την απόδοση και την αυτονομία σε σχέση με τον δίζελ. Άλλο ζήτημα είναι η ασφάλεια. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την ε, εκπόνηση της ε, ανάλυσης αντικτύπου και τις σχέσεις οικονομικής αποδοτικότητας. Έχουμε δει πολύ ανησυχητικά ε, βιντεάκια στο YouTube. Βλέπουμε ένα λεωφορείο των δημόσιων μεταφορών με επιπιεσμένο αέριο το οποίο εκρήγνεται. Πολύ ανησυχητικό και, και μας προβληματίζουν τέτοια περιστατικά. Μας δείχνουν λοιπόν ότι πρέπει να βελτιωθεί η τεχνολογία. Ποιε είναι οι λύσει που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Καλύτερη ενημέρωση από τους κατασκευαστές και τους παρόχους καυσίμου. Ε, καλύτερη πρόσβαση και πιο εύκολη πρόσβαση στην, στα κεφάλαια επενδύσεων. Εχέγγυα για τις επαρκείς ε, επιστροφές και απόσβεση της επένδυσης, ε, αποζημίωση για ενδεχόμενη λύση της μείωση της ικανότητας μεταφοράς και ούτω καθεξής. Άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν να, να αξιοποιηθούν όλες αυτές τις εναλλακτικές για όλες τις μορφές μεταφορών. Το υδρογόνο και η ηλεκτρική ενέργεια, για παράδειγμα, στις ε, μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις και το πεπιεσμένο για τις μεγάλες αποστάσεις. Πρέπει να γίνει περισσότερη έρευνα για να δούμε πώς αυτά τα αναλεκτικά καύσιμα μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλες τις ε, μορφές ε, οδικών μεταφορών. Υπάρχουν κάποιες ε, ενδιαφέρουσες δοκιμές στη Γερμανία με κάποια ε, φορτηγά ε, με την οποία εκπονεί η Siemens με στήριξη και της γερμανικής κυβέρνησης. Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Χρηματοδότηση τώρα. Ποιο είναι το κόστος και μπορούμε να διατηρήσουμε αυτό το κόστος σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Ποιος θα αναλάβει το κόστος και με ποιον τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν διάφορες ε, λύσεις εδώ, ε, τα έσοδα των κρατών μελών από τους ε, φόρους, υπάρχει υπάρχουν πολλές λύσεις. Μετά έχουμε τη βιομηχανία. 26 δις ακούσαμε επενδύει ο κλάδος πάροχοι υποδομών και ο τελικός χρήστης. Είναι σημαντικό κυρίε και κύριοι πάντα ο καθένας να, αναλαμβάνει και ένα ε, δίκαιο τμήμα των κερδών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώσατε και στην ώρα σας. Στη συνέχεια έχουμε τον κύριο Ομπέρτο Γκουίντα, ο οποίος είναι διευθυντής από την UITP και από ό,τι κατάλαβα εσείς είστε αυτού που έχετε τα οχήματα που εκρήγνεται. Έξι λεπτά. Δεν εξαιρέγει αυτό το λεωφορείο, αλλά είχε πιάσει φωτιά όντω στη μία του πλευρά και αρκετά μεγάλη. Δύο λόγια λοιπόν για την UATP καταρχάς. Η UATP είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Δημοσίων Μεταφορών. Εκπροσωπούμε 3.400 ε, μέλη από 90 χώρες, επομένως είμαστε ένας πολύ μεγάλος παγκόσμιος οργανισμός και περιλαμβάνουμε και όλους τους ενδιαφερομένους ε, δημοσίων μεταφορών από τη βιομηχανία, από προμηθευτές ε, μέχρι και διάφορους διαχειριστές ε, αλλά και πανεπιστήμια και ερευνητικά εργαστήρια. Κάποια βασικά στοιχεία για την καθαρή ενέργεια και τις δημόσιες μεταφορές διότι είναι βασικό στοιχείο και υπάρχουν και συγκεκριμένες προκλήσεις περικινητικότητας. Κάθε χρόνο έχουμε 60 δισεκατομμύρια μεταφορών που γίνονται σε οδικά δίκτυα, λεωφορεία αλλά και σιδηροδρόμους ε, σε περιφερειακό επίπεδο. Άνω του 100% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η οικονομική αξία των δημοσίων υπηρεσιών ε, στις μεταφορές και δημιουργούνται 1,2 δισεκατομμύρια ε, άμεσες θέσεις εργασίας για να μην υπολογίσουμε και τις έμεσες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται. Προσπαθούμε να επιτύχουμε τους βασικούς στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής που εντοπίζονται στην Λευκή Βίβλο, δηλαδή ε, να μην υπάρχει ε, χρήση άνθρακα στις δημόσιες μεταφορές και προσπαθούμε να επιτύχουμε το στόχο αυτό και θέλουμε να βοηθήσουμε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Κύριε Γουίντε, καταλαβαίνω ότι 6 λεπτά είναι ε, λίγος χρόνος, αλλά μήπως θα μπορούσατε να μιλάτε λίγο πιο αργά, διότι δεν σας προλαβαίνω διερμηνείς. Ναι, ζητώ συγγνώμη. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να έχουμε και νέα γενεά ε, λεωφορείων και ε, Πολλά από τα περιφερειακά συστήματα ήδη είναι ηλεκτρικά, ηλεκτροκινητά, έχουμε ηλεκτρικά λεωφορεία τα οποία χρησιμοποιούνται σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Σήμερα λοιπόν υπάρχει ένα μερίδιο που είναι ήδη στο 50% της ηλεκτρικής ενέργειας και προβλέπουμε να ε, επιτύχουμε περαιτέρω χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους και μπορούμε να το επιτύχουμε είτε μέσω ηλεκτρικής χρήσης ε, του συστήματός μας, και παρά το γεγονός ότι σήμερα το συνολικό κόστος ε, δεν ε, ε, κάνει ελκυστικές αυτές τις υποδομές. Γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζουμε και την πρόταση οδηγίας ε, για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων και κυρίως καλωσορίζουμε και την προσέγγιση να εξετάσουμε όχι μόνο τα οχήματα αλλά να αναπτυχθεί και κατάλληλη υποδομή. Και θεωρούμε ότι η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όχι μόνο για τον εξηλεκτρισμό αλλά και για άλλα θέματα τα οποία αφορούν την ε, κινητικότητα. Στη διάρκεια του περασμένου έτους, οι πολιτικές συζητήσεις για τα εναλλακτικά καύσιμα και την ηλεκτρική, και η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές ε, αφορούσε την εισαγωγή ηλεκτρικών οχημάτων. Αλλά όπως έλεγε παλιά ο πρώην Γενικός Διευθυντής μας, ε, ε, συμφόρηση με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ναι μεν είναι καθαρή, δεν παράγονται ε, εκπομπές ρήπων, αλλά εξακολουθεί να είναι συμφόρηση. Προσπαθούμε λοιπόν να χρησιμοποιούμε τα δημόσια μέσα μεταφορές για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις προκλήσεις που υπάρχουν και στις αστικές αλλά και στις υπαίθριες περιοχές και θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα μεταφορών που ήδη σήμερα έχει πολύ ε, χαμηλή χρήση άνθρακα και αυτό θα μας βοηθήσει να έχουμε και συνδυασμένες μεταφορές με ηλεκτρική ενέργεια. Και να σας πω ότι η βασική ε, μορφή ηλεκτρικής κινητικότητας προέρχεται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ένα από τα βασικά στοιχεία για να αναπτύξουμε αυτές τις κρίσιμες υποδομές βέβαια είναι το κόστος. Ιδίω σε καιρό που υπάρχει έλλειψη πόρων και είναι ε, περιορισμένοι προπολογισμοί. Έχουμε όμω και κάποια στοιχεία τα οποία μα δείχνουν τι έχουμε ήδη όσον αφορά τι ηλεκτρικέ εγκαταστάσεις. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτέ και να μην δημιουργήσουμε νέε υποδομέ. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τι ήδη υπάρχουσε ε, ε, δομές των δημοσίων μεταφορών και να χρησιμοποιηθούν αυτά ως υποσταθμοί. Έχουμε δυνατότητα λοιπόν για διευκόλυνση ε, συνδυασμένων μεταφορών μέσω της χρήσης αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας. Η Γερμανική Ένωση Δημοσίων Μεταφορών έκανε μια σχετική μελέτη και αναλύσαμε και την έννοια που έχουμε εδώ στη διαφάνεια για να χρησιμοποιούνται ε, συστήματα ε, ηλεκτρικών ε, μεταφορών ε, μέσω αυτών των υποσταθμών για να μπορούμε να έχουμε σημεία επαναφόρτησης εκεί. Και υποστηρίζουμε αυτό το οποίο σχολιάστηκε και από την ε, πλατφόρμα για την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας των μεταφορών μέσω δυνατότητας συνδυασμένων μεταφορών στις δημόσιες μεταφορές. Και κάτι τελευταίο για να ολοκληρώσω. Όπως σας είπαμε, η προσέγγιση αυτή είναι μια προσέγγιση που θεωρούμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα θέματα και όχι μόνο στις υποδομές. Το να υπάρχουν συγκεκριμένε υποδομές ε, και μέτρα διαχείρισης της κίνησης ε, για να αυξήσουμε την ε, εμπορική ταχύτητα έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ αποτελεσματικά. Θα πρέπει να υπάρχουν λεωφοριολορίδες για να υπάρχουν πιο ελκυστικές υπηρεσίες διότι έτσι έχουμε 20% λιγότερο κατανάλωση όπως έχει αποδειχθεί και αυτό θα μπορούσε να σημαίνει και ότι έχουμε 20% λιγότερες εκπομπές. Αυτά από πλευρά μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάουν από το Πόλες. Ο κύριος Χάουν από το Σας ευχαριστώ που μας προσκαλείτε σε αυτή την ακρόαση. Είμαστε μια ένωση πόλεων και περιφερειών από 17 χώρες και θέλουμε να υποστηρίξουμε τα μέλη μας στο να βρουν καινοτόμες λύσεις για ένα βιώσιμο σύστημα κινητικότητας σε, στις πόλεις και στις περιφέρειες. Αυτό περιλαμβάνει και την ηλεκτροκινητικότητα που αναφέρατε. Είμαστε τμήματα αυτής της ε, ε, πλατφόρμας καινοτομία που παρουσίασε και ο κύριος Κρίστη προηγουμένως. Δεν είμαστε εναντίον τη προσέγγισης τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Αντίθετα, εργαζόμαστε μαζί της, αλλά εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία στην ηλεκτροκινητικότητα. Και μα ενδιαφέρει το να μπορούμε να έχουμε μια υποδομή επαναφορτισμού. Πέντε κύρια σημεία θέλω να τονίσω. εμεί χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρξει μια υποδομή επαναφόρτησης. Δίνουμε λοιπόν να πρέπει να δώσουμε ένα σωστό μήνυμα προς την αγορά. Δεύτερον, πιστεύουμε ότι η μετάβαση προς μια μορφή μεταφοράς με ηλεκτρικό, ηλεκτρική ενέργεια και η εισαγωγή των οχημάτων θα πρέπει να είναι τμήμα μιας στρατηγικής για μια πιο βιώσιμη μορφή μεταφορών. Δεν θέλουμε ηλεκτροκινητικότητα απλώ και μόνο αφεαυτής. Θέλουμε μια πιο βιώσιμη μορφή μεταφορών στις πόλεις και στις περιφερειές μας. Πρέπει να παίξει φυσικά η ηλεκτροκινητικότητα κάποιο ρόλο σε όλα αυτά. Μπορεί να παίξει και καταλητικό ρόλο για τη μετάβαση προς ένα βιώσιμο σύστημα μεταφορών. Θεωρούμε λοιπόν ότι το πλαίσιο αυτό δράσης σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να περιλαμβάνει και μια και για την εισαγωγή της ηλεκτροκινητικότητας σε αστικό και περιφερειακό επίπεδο. Και επομένως αυτό θα πρέπει να έχει ως στοιχείο και μια υποδομή για επαναφόρτιση οχημάτων. Και έτσι αυτό σημαίνει και μια πιο ολοκληρωμένη διαχείριση ενέργειας. Υποστηρίζουμε στόχους για το 2020 για το ποσοστό ε, σημείων επαναφόρτησης και την ελάχιστη απόστασή τους, όλα αυτά θα πρέπει να αποφασιστούν σε ένα εθνικό πλαίσιο. Και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις ποικιλομορφίε των κρατών μελών. Μπορεί σε ορισμένε περιοχές να μην χρειαζόμαστε ε, τόσα σημεία επαναφόρτησης, τουλάχιστον δείχνουν οι επιδείξεις που έχουμε κάνει με οχήματα, ενώ σε άλλες περιοχές είναι πολύ πιο υψηλό το ποσοστό των σταθμών που χρειάζεται. Αν λοιπόν έχουμε μεγαλύτερη ευκαμψία στα κάτι μέλη σε σχέση με τους σταθμούς επαναφόρτησης, μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ε, αποδοτικότητα. Επίσης το θέμα των ε, υποδοχέων των πριζών υπαριθμών της κατηγορίας 1 και 2. Εδώ θα πρέπει να βρούμε μια λύση η οποία επιτρέπει και τα παλαιά οχήματα να μπορούν να επαναφορτίζονται σε όλη την Ευρώπη. Και το τελευταίο σημείο το οποίο θέλω να δείξω είναι ότι εμεί θέλουμε να έχουμε και την υποστήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας για να υπάρξει μια υποδομή επαναφόρτιση. Αυτό μπορεί να αποτελέσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική γιατί θα μπορέσει να βοηθήσει τις στρατηγικές προς την ηλεκτροκίνηση. Θα πρέπει όμως να υπάρξει σωστός συντονισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών ε, οργάνων, να υπάρξει και κατάλληλη χρηματοδότηση και όλα αυτά θα πρέπει να μεταλαμπαδεύονται υπό μορφή πληροφόρησης προς πολίτες από ενιαίους φορείς με κοινούς μηχανισμούς και έτσι θα μπορούσε να υπάρχει μια υποστήριξη από την Ευρώπη με κάποιο παρατηρητήριο για την βιώσιμη κίνηση. Και αυτά λοιπόν από την παρουσίασή μου. Έρχομαι μονάχα στην τελευταία διαφάνεια που αναφέρεται στο σχέδιο TIDE Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να πάρει τα απαραίτητα μέτρα που έχουν να κάνουν με την διαλειτουργικότητα και εμείς θέλουμε να καθορίσουμε τους τρόπους με τους οποίους θα χρηματοδοτηθούν οι σταθμοί επαναφόρτισης. Όλα αυτά θα είναι εξαιρετικά σημαντικά και συναρπαστικά αν τεθεί σε εφαρμογή αυτή η οδηγία με μορφή παρά κοντά σε αυτή που έχει τώρα. Ευχαριστώ ο κύριος Μαρτίνες Μάρτες από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω σύντομα κάποιες παρατηρήσεις ε, για τον τομέα των χρυσών μεταφορών και για τη χρηματοδότηση αυτού του κλάδου που αναφέρθηκε πολλές φορές από προηγούμενες ε, ομιλίες και τις ε, προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ως Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γι' αυτό ε, συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε σε δραστηριότητε που θα έχουν τον μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές πολιτικές και του πολιτικούς μας στόχους. Από του βασικού στόχου είναι οι βιώσιμε βιώσιμες και η κλιματική αλλαγή. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λιγότερη ενέργεια και καθαρότερη ενέργεια για να μειώσουμε τον αντικό αντίκτυπο ε, στο περιβάλλον. Γι' αυτό η ανάπτυξη μια ενιαία αγορά για τι ε, εναλλακτικέ υποδομέ ε, υποδομές εναρκτικών καυσίμων και αντίστοιχων οχημάτων βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής μας. Και η ανάπτυξη του δικτύου TNT είναι κύριος στόχος. Και μάλιστα μόνο το 2011 δαπανίσαμε ε, δις ευρώ σε αυτόν τον κλάδο. Και είναι κάτι που στηρίζει η τράπεζά μας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε επενδύσει πάνω από 70 δις στον τομέα των μεταφορών. και το μερίδιο των, της χρηματοδότησης προς δομέα φορών είναι περίπου 25% όλης της, της ε, δανειοδότησης της τράπεζάς μας. Όμως ε, έχουν αλλάξει κάποια στοιχεία, ιδίως σε ό,τι αφορά ε, τα προγράμματα των χερσαίων μεταφορών που έχουν αυξηθεί την τελευταία δεκαετία και έχουμε δει αύξηση της δανειοδότησης και προς τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων παρότι είναι λίγες οι ε, τέτοιες προσπάθειες. Να μιλήσω λίγο για τη χρηματοδότηση, τα τρία βασικά μας ε, εργαλεία. Πρώτο, είναι η τεχνική συνδρομή. Συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε ε, δυνατότητες να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να προετοιμάσουν ε, προγράμματα που μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση. Το RSFF βελτιώνει την πρόσβαση στη δανειοδότηση για τέτοια προγράμματα που αφορούν τέτοιες υποδομές εναλλακτικών καυσίμων και η πρωτοβουλία Ελένα δίνει χρηματοδοτική ενίσχυση και συνδρομή για συγκεκριμένες επιχειρηματικές προσπάθειες στον τομέα των εναλλακτικών καυσίμων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η πρωτοβουλία Jaspers βοηθά τα νέα και μελλοντικά κρατημέλη να ε, εκπονήσουν τέτοιε επιχειρηματικέ προσπάθειε. Όλα αυτά τα προγράμματα λοιπόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση μελλοντικών ε, προσπαθειών στον τομέα αυτό. Δεύτερο, είναι η παραδοσιακή χρηματοδοτική και δανειοδοτική μας δραστηριότητα που είναι βασική μας ε, δραστηριότητα. 90% των ε, οικονομικών μας δεσμεύσεων αφορούν την δανειοδότηση. Και η στήριξή μας είναι πολλές φορές κεντρική σημασία για την προσέλκυση άλλων επενδυτών. Βεβαίως η συνέχεια αυτής της προσπάθειας απαιτεί μια πολυτομιακή προσέγγιση και εμείς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε πολλούς ε, διαφορετικούς φορείς όπως είναι ε, διάφορες επιχειρήσεις, κατασκευαστικές και το Τέλος έχουμε μια πληθώρα οικονομικών και χρηματοοικονομικών μέσων. Το ΙΠΕΚ έχει συσταθεί για την ανάπτυξη του δημόσιου τομέα κατά την ε, εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων και εταιρικών σχέσεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Τέτοια προγράμματα λοιπόν που θέλουν να αναπτύξουν προγράμματα αναλλακτικών καυσίμων στο TNT μπορούν να αξιοποιήσουν και το λεγόμενο LTGG. Κλείνοντας, ήθελα να πω ότι έχουμε πολλά, έχεις πολύ σύγχρονα εργαλεία για την χρηματοδότηση ε, μακροπρόθεσμων ε, προγραμμάτων. Βεβαίως η ανάπτυξη αυτού του τομέα δεν θα είναι εύκολη με δεδομένης και της οικονομικής συγκυρίας. Απαιτείται και ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών. Εμείς βεβαίως είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε τις ε, τυχόν, όποιες προσπάθειες και πρέπει να φέρουμε αυτές τις προσπάθειες ε, στο επόμενο τους ε, στάδιο και αν καταφέρουμε να καταστήσουμε τις μεταφορές ε, πιο βιώσιμες και καθαρές, αυτό θα ωφελήσει όχι μόνο τα ενδιαφερόμενα μέλη αλλά και εν γέννη για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ευχαριστώ. Εκτός από τον κύριο Φιντάντσα, ποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο για τα θέματα αυτά. Κυρία Λίχτεμπέργκεν, Ρικέ, Ντεπάκερ. Ωραία λοιπόν. Κύριε Φιντάντσα, τρία λεπτά και όλοι οι υπόλοιποι από δύο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή τη φορά δεν έχω πολλές ερωτήσεις. Μία παρατήρηση και μετά ε, κάτι συγκεκριμένο. Τελικά έχω και μια ερώτηση. Στην τελευταία παρέμβαση του κυρίου Μάρτενς μου δόθηκε εντύπωση ότι όσον αφορά τη χρηματοδότηση και μην το πάρετε στραβά, το λέω με πάσα συμπάθεια, ε, υπεκφεύγεται λίγο. Θα ήθελα να σας ε, πω λίγο την άποψή μου, την άποψη που επικρατεί εδώ στην Επιτροπή μας και την οποία θα αναπτύξουμε και στην ε, διάρκεια της έκθεσης. Έχουμε δύο ουσιαστικά προβλήματα. Το ένα αφορά τις ε, χρηματοδοτήσεις. Ε, υπάρχουν πολλές δυσκολίες για το ποιο πληρώνει και δεύτερον υπάρχει και το θέμα των στόχων. Μπορούν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι το 2020 είναι συμβατά με την κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή στην αγορά και την κατάσταση που έχουμε στα διάφορα κράτη-μέλη και στις διάφορες περιοχές. Και πρέπει να επικεντρωθούμε κατά προτεραιότητα σε αυτές τις πτυχές για να διασκεδάσουμε κάποιες αμφιβολίες και να κάμψουμε και κάποιες αντιστάσεις που υπάρχουν και στο εσωτερικό της Επιτροπής μας, αλλά ε, που μας περιμένουν και στις διαπραγματεύσεις στη συνέχεια με το Συμβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν σε ένα σύντομο δεύτερο γύρο να διευκρινίσετε λίγο καλύτερα αυτές τις δύο πτυχές, διότι έτσι μπορούμε να έχουμε πολύ περισσότερα επιχειρήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Και ε, εδώ θα ήθελα και κάποια παραδείγματα για βέλτιστες πρακτικές, παραδείγματα τα οποία έλαβαν χρηματοδότηση χωρίς ε, υπερβολική χρήση δημοσίων κονδυλίων, αλλά με άλλους τρόπους, όπως για παράδειγμα φορολογικά κίνητρα, διάθεση δημόσιων χώρων για εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού ή επαναφόρτησης, ε, προβλέψεις ε, σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και δημόσιες συμβάσεις ε, συγκεκριμένων προδιαγραφών για τις προϋποθέσεις επαναφόρτησης. Δηλαδή, να πάμε προς μια κατεύθυνση ώστε να ε, δείξουμε πώς μπορούν να μειωθούν στο ελάχιστο οι δημόσιες επενδύσεις για να μπορέσει όμως ταυτόχρονα να υλοποιηθεί και αυτό και το σχέδιο. Μια συγκεκριμένη ερώτηση όμως προς τον κύριο Λάρος. Το πού θα τοποθετούνται οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Εσείς θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο όπως προβλέπετε κάθε λιμένες, ε, λιμένας να μην περάσουμε στα εσωτερικά ύδατα, να δούμε μόνο τους θαλάσσιους λιμένες. Πρέπει να διαθέτει όπως προβλέπετε και μια εγκατάσταση αποθήκευσης και διαμονωμής ή θεωρείτε ότι θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη και να επιλέξουν αυτά που θα έχουν τους σταθμούς. Η κυρία Λιχτεμπέργκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα ερώτημα για τις ε, πόλεις. <coughs> κυρία, Χάουν. Όταν μιλήσατε για το κόστος το οποίο προκύπτει όταν σε κάποια γειτονιά θέλουμε να έχουμε υποδομές ή αν έχουμε κάποιο κεντρικό χώρο υποδομών για την ηλεκτροκινητικότητα. Πώς γίνεται η εκτίμηση του κόστους. Έχετε κάποια μοντέλα τα οποία μπορούν να μας επιτρέψουν να κάνουμε κάποια εκτίμηση της, ε, ε του κόσμου προκύπτει. Τώρα χωριστά από τα μοντέλα για το car sharing, για, το, για την αποκοινού χρησιμοποίηση των αυτοκινήτων. Ένα δεύτερο ερώτημα το οποίο θέλω να θέσω. Είναι δυνατόν να επιληθεί το πρόβλημα αυτό το οποίο θα αποκύψει με την έλλειψη χώρου για τις υποδομές θα γίνει με εταιρικε σχέσει δημόσιου δημόσιο-ιδιωτικού τομέα και τι γίνεται για την ε, μεγαλύτερη προσέλκυση αυτών που χρησιμοποιούν το δικό τους ε, αυτοκίνητο. Μήπως θα πρέπει να υπάρχει μια προσέλκυση αυτών στις δημόσιες μεταφορές και να υπάρξει μια αλλαγή των δομών. Και στον κύριο Γκουίντα τώρα θέτω ένα ερώτημα. Αν υπάρχει μια εμπειρία για το κόστος, την διάρθρωση του κόστους που προκύπτει από την ε, μετάβαση σε αυτές τις μορφές κίνησης. Ποιος είναι αυτός ο οποίος επιφορτίζεται το κόστος για το συνολικό κόστος στη διάρκεια ζωής μιας μπαταρίας, παραδείγματος χάρη. Είναι χωριστά απόβλητα, είναι ειδικά απόβλητα, πρέπει να αντιμετωπιστούν με ένα ειδικό τρόπο Πώς ενσωματώνεται αυτό το κόστος μιας μπαταρίας ηλεκτρικού οχήματος. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη ακόμα και αν έχουμε μεγαλύτερη μεγαλύτερα κίνητρα για τη χρήση των δημοσίων μεταφορών παραμένει το κόστος για τη χρήση παραδείγματος χάρη των μπαταριών για την ε, ανακύκλωσή τους, για την τελική εναπόθεση των αποβλήτων κτλ. Έχετε κάποιο μοντέλο για όλα αυτά, ο κύριος σας ευχαριστώ. <clears throat> Δύο ερωτήματα έχω να θέσω στον κύριο Λάρος καταρχήν. Με έκπληξη σας άκουσα να μιλάτε για τις εναλλακτικέ ενέργειες στο θαλάσσιο τομέα χωρίς να αναφέρεστε στο θέμα της μείωσης της επιβολής μείωσης των εκπομπών θείου που οξυδιών του θείου που θέτει ένα μεγάλο πρόβλημα για τις θαλάσσιες μεταφορές που χρησιμοποιούν παραδοσιακά καύσιμα. Επομένω υπάρχουν ιδιαίτεροι περιορισμοί για το θαλάσσιο χώρο. Επίσης αναφερθήκατε στο γεγονός ότι το φυσικό αέριο, <coughs> το υγροποιημένο φυσικό αέριο καλύπτει τόσο μεγάλο μέρος του όγκου των πλοίων που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλες αποστάσεις. Γιατί εγώ ήμουν παρόν σε μία συνδιάσκεψη για τα θέματα αυτά με εμπειρογνώμονες για τα θέματα αυτά και δεν είπε κανένας λέξη για αυτό το θέμα. Ιδίως όταν μιλάμε για πλοία ωκεανοπόρα που πηγαίνουν στα μεγάλα λιμάνια που μεταφέρουν ε, φυσικό αέριο σε μεγάλες αποστάσεις, κανείς δεν αναφέρθηκε σε αυτό το ερώτημα. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πόσο χώρο καταλαμβάνει η αποθήκευση του φυσικού αερίου σε ένα πλοίο, πόσο περισσότερο από ότι αν έχουμε ένα φυσιολογικό, ένα συμβατικό καύσιμο και αν αυτό από μόνο του οδηγεί σε περιορισμούς για τη χρήση του, αερίου, γιατί φυσικά εμποδίζει την μεταφορά ωφέλιμου φορτίου. Εγώ δεν έχω ακούσει αυτή την προβληματική στο παρελθόν. Και ένα ερώτημα που στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Στο πλαίσιο του Connecting Europe έχουμε ε, δίκτυα μεταφορών αλλά έχουμε <clears throat> και δίκτυα ενέργειας. Και μπορεί να προκύψει μια συνέργεια μεταξύ των δύο δικτύων γιατί μας ενδιαφέρει η μεταφορά της ενέργειας αλλά μας ενδιαφέρει και η χρήση ενέργειας για, την, για τις καθαρές μεταφορών. Δεν βλέπω το Συμβούλιο να έχει ενδιαφερθεί πάρα πολύ για το θέμα αυτό και δεν υπάρχει ευρεία συζήτηση για τα θέματα αυτά. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να ενδιαφέρει περισσότερο την αγορά να εξασφαλίσει τις συνέργειες αυτές. Γιατί τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία σε τέτοιου είδους επενδύσεις και τότε και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Τα έχει διερευνήσει αυτά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα, χρηματοδοτήσει για την ανάπτυξη νέων δικτύων. Κύριο Στεμπάκερ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ε, εξηγήσεις που μας δώσετε. Έχω κάποια ερωτήματα. Κάτι το οποίο καθίστε το λένε και πιο σαφές είναι ότι ολόκληρο το δίκτυο μεταφορών ε, λειτουργεί όλα είναι και πιο συστημικά. Ε, δηλαδή δεν είναι μόνο τα κάψιμα, είναι και υποδομές, είναι και τα οχήματα, όλα μαζί. Το βασικό ερώτημα λοιπόν είναι, ακούσαμε πολλά για το τι μπορεί να κάνει ο δημόσιος τομέας, αλλά οι ιδιωτικοί φορεί πώ θα συμμετάσχουν. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Πριν από δύο εβδομάδε, μια εταιρεία που έχουμε ε, χρησιμοποιήσει πολλέ φορέ εδώ ω παράδειγμα ε, για τι ε, επενδύσει των ιδιωτικών φορέων, χρεοκόπησε. Πώ λοιπόν μπορείτε να δώσετε εχέγγυα ότι και οι ιδιωτικοί φορεί ε, που μπορούν να επενδύσουν ε, θα τα καταφέρουν. Γιατί κατά τη γνώμη μου αυτό δεν έχει αναφερθεί αρκετά σε αυτή τη συζήτηση. Δεύτερον, αν υπάρχει τέτοια, τέτοιο ενδιαφέρον και επένδυση από τον δημόσιο τομέα, αυτό πρέπει να γίνεται και με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο. Εμεί ω κυβερνήσει φανήκαμε. Ε, στην επιλογή των νικητών και όχι των χαμένων. Μπορούμε λοιπόν να επενδύσουμε σε κάθε τεχνολογία. Όχι, πρέπει να κάνουμε μια επιλογή. Αλλά αν κάνουμε μια επιλογή μπορεί να χάσουμε ευκαιρίες σε άλλες τεχνολογίες. Πώς μπορούμε λοιπόν να μεριμνήσουμε για αυτό το στοιχείο. Και τέλος, για ε, τις θαλάσσιες μεταφορές, ήδη ο συνάδελφος τα ανέφερε. Υπάρχει το ζήτημα των νέων περιβαλλοντικών περιφερειών που πρέπει να ε, εφαρμοστούν μέχρι το 2015, αν δεν κάνω λάθος, και αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο στους στόλους. Πολλά λέγονται για επενδύσεις ε, στην παράκτητα πλευρά, αλλά τι θα γίνει για την ανανέωση του στόλου. Όλα αυτά τα σκάφη θα πρέπει ε, με κάποιον τρόπο να ανανεωθούν ή να αναπαλαιωθούν. Πώς θα συμβάλλει ο ιδιωτικό τομέα λοιπόν σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε και πάλι το λόγο στο πάνελ για να απαντήσει εν συντομία. Επαναλαμβάνω ότι αν δεν, έχετε, δεν σας φτάνουν τα δύο λεπτά για να απαντήσετε, μπορείτε να στείλετε τις απαντήσεις σας γραπτός. Ο κύριος Λάρους το λόγο. Πρώτον, για τον όγκο ή τη χωρητικότητα. για το υγροποιημένο. μεταφέρεται στους μειών 160 βαθμούς. Άρα χρειαζόμαστε και ε, μια μονομένη εγκατάσταση αποθήκευσης και οι προϋποθέσεις ασφαλείας, όπως έχουν τώρα τουλάχιστον, είναι πολύ αυστηρότερες σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο έκρηξης. Και έτσι η δεξαμενή είναι το καλύτερο περιβάλλον αποθήκευσης. Αυτό έχουν ως αποτέλεσμα ότι σε σύγκριση με το βαρύ, ε, το βαρύ αργό πετρέλαιο χρειαζόμαστε πενταπλάσιο χώρο για την ε, αποθήκευση του αερίου. Υπάρχει λοιπόν σοβαρό πρόβλημα. Όπως είπα και προηγουμένως, αν υπάρχει δυνατότητα συχνότερων εφοδιασμού, τότε διευκολύνουν τα πράγματα. Έχουμε συζητήσει τη δυνατότητα αξιοποίηση ε, του φυσικού αερίου ως καυσίμου και τροποποίηση των περισσότερων ε, μηχανών για την ε, χρήση του υγροποιημένου φυσικού Τα λεγόμενα scrubber ε, αξιοποιούνται όταν έχουμε ε, καύσιμο χαμηλής ποιότητας και θέλουμε εκεί να, ε, να πληρούμε και τις προεταγραφές ΙΚΑ. Εκεί είτε παίρνουμε πολύ καθαρά κάψιμα, είτε ε, επενδύουμε σε άλλες μεθόδους. Τώρα, για την δυνατότητα αποθήκευσης, θεωρώ ότι όλα τα μεγάλα λιμάνια στην Ευρώπη πρέπει να έχουν μια μορφή αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου. Εντάξει, βέβαια είναι υπερβολικό να ζητήσουμε ότι κάθε λιμάνι στο Ρήνο θα έχει τη δική του εγκατάσταση. Όμως είναι ζήτημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει λοιπόν αυτή η αγορά να λειτουργήσει, να επιλέξει του δικού τους ε, σταθμού αναφοδιασμού. Κύριος Πηλιέ, ευχαριστώ. Ορισμένε παρατηρήσει. Πρώτον, για, τις, για του στόχου. Από μα είμαστε υπέρ φιλόδοξων στόχων. Οι μη φιλόδοξοι στόχοι ενδεχομένω να αναβάλουν όλη αυτή την ιστορία. Και είναι κάτι απαραίτητο. Ήταν απαραίτητο και πριν από 10 χρόνια, είναι απαραίτητο και τώρα, το στομότερο δυνατόν. Γιατί πρέπει να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μα ίχνος για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Οι εταίροι αυτού του ιδιωτικού τομέα ήδη συμμετέχουν, όμως πράγματι από πλευράς ε, εμπορευομένων στις μεταφορές πρέπει να συμμετέχουν ε, σε μεγαλύτερο βαθμό ε, στην έρευνα, ιδίως σε ό,τι αφορά τις δοκιμές και οι κατασκευαστές οχημάτων και η παραγωγή καυσίμων θα πρέπει να εξετάσουν τη βιωσιμότητα και να βρίσκουν λύσεις σε ε, αρχικό επίπεδο. Κατά πόσο τώρα είναι βαρχιπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο. Τα εξετάσαμε και ε, με την αντίστοιχη ομάδα εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι έλεγχοι που, κίνδυνοι που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Είναι ένα ρίσκο που θα πρέπει να αναλάβουμε γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλη εναλλακτική λύση που μπορεί να αντικαταστήσει πλήρω το πετρέλαιο. Αν ε, υιοθετήσουμε αποφάσεις πολύ γρήγορα, μπορεί να χάσουμε ε, και τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Γι' αυτό πρέπει να επενδύσουμε σε δοκιμές, δοκιμές ελέγχους και ελέγχους. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Γκουίντα. Καταρχάς, όσον αφορά τους στόχους από πλευράς δημοσίων μεταφορών, ο στόχος μας ετέθη σε σχέση με το μερίδιο της αγοράς. Ήταν πολύ ευρύτερος λοιπόν από τη συγκεκριμένη έννοια της ηλεκτρικής κινητικότητας και το καθεξής. Ο στόχος του διπλασιασμού λοιπόν του μεριδίου της αγοράς το 2025 είναι αυτός που μας απασχολεί. Όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές, βεβαίως αυτό έχει σχέση ε, και έχουμε κάποια παραδείγματα που... Ε, είναι ανάλογα με τη χώρα, ε, μπορούμε να σας δώσουμε τέτοιες πληροφορίες ε, με περισσότερες λεπτομέρειες ε, γραπτός. Το ίδιο όσον αφορά το κόστος του κύκλου ζωής και σε γενικές γραμμές για την ανάλυση will-to-will. -will. Υπάρχουν υπαρχουν έρευνες ανάλογα με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τις μπαταρίες. Υπάρχουν κάποιες ύλες οι οποίες πρέπει να προέρχονται από συγκεκριμένε χώρες σε κάποιες περιπτώσεις ε, ορισμένες φορές δεν είναι λύση λοιπόν του προβλήματος, αλλά μετατόπιση του προβλήματος από το μία πλευρά στην άλλη. Και έχουν γίνει και κάποιες μελέτες από πλευράς κόστους και νομίζω ότι και εδώ θα μπορούσα να ζητήσω από τους εμπειρογνώμονές μου να σας δώσουν κάποιες περαιτέρω πληροφορίες. Τώρα, όσον αφορά την ε, ουδετερότητα της τεχνολογίας, ε, βεβαίως και εμείς ενδιαφερόμαστε για την ουδετερότητα της ε, τεχνολογίας. Σήμερα υπάρχει μια νέα γενιά λεωφορείων που κινούνται με δίζελ, που είναι και θα εξακολουθήσουν να είναι η ραχοκοκαλιά των δημοσίων μεταφορών για τα επόμενα χρόνια. Είναι πιο καθαρά και έχουν και καλύτερη απόδοση από περιβαλλοντική σκοπιά, κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει εξίσου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω και στον κύριο Φιντάντσα και στην κυρία Λιχτεμπέργκερ ταυτόχρονα, διότι θεωρώ ότι είναι αντίστοιχε οι ερωτήσει ε, για την οικονομική κατάσταση και τι οικονομικέ προποθέσει. Το ερώτημα είναι ποιο πληρώνει και αν έχουμε και τα λεφτά να τα πληρώσουμε. Καταρχάς να σας πω ότι εγώ προσωπώ το δημόσιο τομέα. Η πίεση λοιπόν προς τα δημόσια οικονομικά υπάρχει και υπάρχουν και πάρα πολλές αρχές που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Καταρχάς θα πρέπει να υπάρξει μια ένδειξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να μην είναι μεγάλο ε, τμήμα της χρηματοδότησης, μπορεί να είναι μικρότερο το τμήμα της χρηματοδότησης, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια ένδειξη από, τον, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω ε, να είναι και θετική στάση του κ. Ρικέ προς αυτό το θέμα θα υπάρχει κάποια δημόσια επένδυση, σίγουρα θα υπάρχουν ιδιωτικέ επενδύσει, αλλά υπάρχουν πολλέ δυνατότητε σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και υπάρχουν και κάποιε εξ αυτών που είναι ήδη εν σήμερα είτε πρόκειται για σύμπραξη με τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ε, ή με τον ε, ε, χώρους στάθμευσης, επιχειρήσεις που ασχολούνται με αυτά, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν ίσως να διαθέτουν ηλεκτρικά οχήματα στους πελάτες. Ε, που σημαίνει ότι ε, έχουν και σταθμούς επαναφόρτησης και αυτό θα είναι τμήμα της στρατηγικής. Μπορεί να είναι και τμήμα μιας δέσμης μέτρων για τις υπηρεσίες. Μπορεί να έχετε, έχετε κάποιες πόλεις, Άμστερνταμ, Βαρκελόνη, ανέφερα πόλεις οι οποίες είναι πολύ προηγμένες σε αυτά τα θέματα και υπάρχουν διάφοροι τρόποι να δούμε την πλευρά της ε, χρηματοδότησης για τους σταθμούς επαναφόρτησης για τα ηλεκτρικά οχήματα. Ελπίζω να μπορέσουμε να σας ε, δώσουμε και περισσότερες λεπτομέρειες ε, και μια συνολική εικόνα σύντομα για να έχετε και μια εικόνα ε, των, ποσών που νομίζω ότι ενδιαφέρουν όλους. Ευχαριστώ κύριος Μάρτεντς. Σας ευχαριστώ για το θέμα της χρηματοδότησης των υποδομών. Εμείς βέβαια είμαστε τράπεζα και μπορούμε όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να δώσουμε δανειοδότηση και μπορούμε να παίξουμε κάποιο ρόλο έναντι δημοσίων αρχών που πρέπει να χρηματοδοτήσουν αυτές τις επένδυσεις και να τις βοηθήσουμε. Αυτό που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια είναι ότι με τα σχέδια αυτά είναι σχέδια α, αυτών οι οποίοι υιοθετούν πρώιμα μια τεχνολογία και είμαστε ακόμα στις <clears throat> αρχές, στις απαρχές αυτών των ε, προσπαθειών και επομένως τα περισσότερα σχέδια έχουν μια κοινή συμμετοχή δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα η τετερική σχέση μια άλλη δομή. Και είδαμε επίσης για τα ταξί, για τις εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων να κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι οι πρώτες κινήσεις για την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων φυσικά αντιμετωπίζουμε κατά περίπτωση όλες αυτές τις προτάσεις χρηματοδότησης. Εξετάζουμε το αν ευσταθεί σε επίπεδο επιχειρηματικό <clears throat> και πρέπει να εξασφαλίσουμε και ότι επομίζονται ένα μεγάλο μέρος του κινδύνου και οι εμπλεκόμενοι σε αυτά τα σχέδια. Όπως είπα και προηγουμένως, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια εξέλιξη με την πίεση των καταναλωτών, αυτών που αγοράζουν αυτοκίνητα, αυτών που ενδιαφέρονται για τις νέες τεχνολογίες. Αλλά είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο για τον ιδιωτικό τομέα για να μπορέσει να επενδύσει στις υποδομές ένα σαφές πλαίσιο και μια σαφής δομή χρηματοδότησης όπου μπορεί κανείς να, <clears throat> να επομιστεί ένα δίκαιο μέρος του κινδύνου. Αυτά είναι προϋποθέσεις λοιπόν για να προχωρήσουμε αυτά τα σχέδια. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρος. Κύριε Ονίδη, θέλετε να πείτε κάτι. Κύριε Φιντάντς, εσείς θέλετε να πείτε κάτι. Καταληκτικές παρατήρησεις. Soltanto alcune brevi considerazioni. Κάποιες πολύ σύντομες τελικές παρατηρήσεις. Καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές ε, και για αυτό το τμήμα της συζήτησης. Πρέπει να πω ότι σε γενικές γραμμές είναι καλή αποδοχή της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία προφανώς ε, έχει μεν φιλόδοξους στόχους, αλλά θεωρώ ότι όσον αφορά τη γενικότερη τοποθέτηση ε, υπάρχει συνένεση. Και επίσης είναι πολύ σημαντικός και ο τρόπος με τον οποίο θελήσαμε να ε, γίνει αυτή η ακρόαση. Δεν επικεντρωθήκαμε όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έναν τύπο εναλλακτικού καυσίμου και μόνο, αλλά θελήσαμε να εμβαθύνουμε σε διάφορες πτυχές, διότι θεωρώ ότι πρέπει να συνειδητοποιούμε όλοι ότι η εναλλακτική λύση στο πετρέλαιο για τις μεταφορές δεν μπορεί παρά να είναι ε, πληθυντικού αριθμού. Σίγουρα δεν υπάρχει μία μόνον λύση. Είναι πολύ σημαντικό και προέκυψε και από αρκετέ παρεμβάσει ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ολιστική προσέγγιση, δηλαδή να λάβουμε υπόψη τα στοιχεία που αφορούν τους κατασκευαστές, τις δημόσιες ε, υπηρεσίες, ε, τους ε, προμηθευτές φυσικού αερίου ή οποιαδήποτε άλλη μορφή καυσίμου, αλλά είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη και τις ανάγκες των πελατών. Είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση του ποιος έκανε το αυγό ή την κότα. Ε, και δεν υπάρχει αγορέ σε κάποιες φορές λέμε, δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι δεν υπάρχει αγορά αν δεν υπάρχει υποδομή. Πρέπει λοιπόν η οδηγία να πιέσει υπό τη μορφή των υποδομών για να ε, αναπτυχθεί και η αγορά. Δεν ξέρουμε ποιο είναι η κότα ή το αυγό ε, και δίνουμε μια σημαντική όθηση και πρέπει να λάβουμε σίγουρα δεόντως υπόψη και τις ανάγκες του καταναλωτή. Άκουσα πολλά πράγματα για τις συνδυασμένες μεταφορές, οι οποίες σίγουρα συνάδουν με τις πολιτικές μας εν γέννη στον τομέα αυτό. Θα ήθελα να εμβαθύνουμε και στο θέμα της ασφάλειας. Άκουσα από τον κύριο Μπιλιέ ε, μία αναφορά σε κάποια ε, στοιχεία τα οποία αναλυθεύουν πραγματικά με ανησυχούν ιδιαίτερους. Ε, δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κάποιος ότι είναι αληθινά. Δεν ξέρω βέβαια μάλλον ο άλλος ομιλητής δεν συμφωνεί. συμφωνώ όμως στην έκκληση για ασφάλεια. Θα πρέπει να έχουμε ίσως κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία αν όντω υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Εγώ δεν είχα την εντύπωση ότι υπάρχουν τόσο σοβαρά προβλήματα ασφάλειας για το φυσικό αέριο. Για τους στόχους νομίζω ότι ε, σε γενικές γραμμές υπάρχει σύμπνοια ε, για το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχουν στόχοι, θα μπορούσαμε ίσως να σκεφτούμε και κάποια επιπλέον στοιχεία ευελιξίας εδώ και θα πρέπει ε, να υπάρχει στο μέτρο του δυνατού για τη χρηματοδότηση, δημόσια κονδύλια, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ε, χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων, αλλά και φυσικά και η ιδιωτική πτυχή, η οποία αναφέρθηκε επανειλημμένω, διότι χωρίς την συνδρομή της δεν μπορούμε να έχουμε αυτές τις επενδύσεις. Και όσον αφορά την πρόταση εναρμόνιση, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικός στόχος, να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα ένας οδηγός ο οποίος χρησιμοποιεί ηλεκτρικό όχημα να έχει τις ίδιες προδιαγραφές και να υπάρχει μια ενιαία αγορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε μια λύση που θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φιντάντσα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ε, λίγο το χρονοδιάγραμμα που έχουμε καθορίσει για το συγκεκριμένο θέμα. Η παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια θα υπάρχει μια προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών μέχρι την 1η Οκτωβρίου και προβλέπεται ψηφοφορία στην Επιτροπή Μεταφορών στις 14 Νοεμβρίου να ευχαριστήσω ε, το δεύτερο γύρο μιλητών, τους κυρίους Μάρτενς, Γκουίντα, Λάρος, Μπιλιέ και Χάον για τη συνεισφορά τους και φυσικά θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τους ομιλητές στο πρώτο πάνελ, ε, Κρίστη κλπ. κλπ. Ε, σας ευχαριστούμε όλους, ευχαριστούμε και για τη σημερινή σας παρουσία και για τις απόψεις που μας παρουσιάσετε. Θα συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας στις 3. Ευχαριστώ πολύ.